So, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting without a long voting. Um, our first point. Το πρώτο σημείο για, την, για σήμερα το απόγευμα είναι οι δείκτες της μετανάστευσης για το 2015, κοινή δημοσίευση του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε το Γενικό Γραμματέα που θα καθυστερήσει κάπως και θα μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή, αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε την κυρία Πάικ από την DG Home και να ξεκινήσουμε με τη δική σας την παρουσίαση. Και απλώς να θυμίσω ότι αυτή η κοινή δημοσίευση του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πρώτη σύγκριση στοιχείων σε διεθνέ επίπεδο όλων των χωρών του ΟΣΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι κινήσει μεταναστών και των παιδιών του έχουμε. Με 37 δείκτε προγραμμούνται σε μεγάλου τομεί. Απασχόληση, εκπαίδευση και δεξιότητε, κοινωνική εντάξει η συμμετοχή των πολιτών και η κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, δύο ειδικά κεφάλαια αφιερώνονται σε συγκεκριμένε ομάδε. Η πρώτη είναι αυτή των νέων με ε, ιστορικό μεταναστών που είναι ένας συγκριτικός δείκτης για την επιτυχία την αποτυχία της ένταξης. Επίτα το δεύτερο είναι η πίκο τρίτη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ένταξη στις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομίζω ότι τα πορίσματα της ε, μελέτης αυτής θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για την Επιτροπή μας. Κυρία Πάικ. Α, ο Γενικός Γραμματέας έφτασε. Να περιμένουμε. So, then Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον κύριο Άγγελ Γκουρία, Γενικό Διευθυντή του ΟΣΑ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεση που μόλις ανέφερα, την έκθεση του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Γκουρία, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μπορώ να σας παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα της νέας μας έκθεσης δείκτες ολοκλήρωσης ε, ή μάλλον ένταξης των μεταναστών για το 2015. Αυτό το έντυπο που σας δείχνω. Ελπίζω να έχετε όλοι αντίγραφα. Αλλά σίγουρα μπορείτε να διαβάσετε και τα σχετικά στην ιστοσελίδα μας. Πρόκειται για μια δημοσίευση που ουσιαστικά είναι μια πρώτη διεθνής σύγκριση σε όλες τις χώρες της Ένωσης και του ΟΣΑ για τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τους μετανάστες και τα παιδιά τους στις χώρες υποδοχής περιλαμβάνει μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο συμπίλημα πληροφοριών για τα ζητήματα της ένταξης. Είναι το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα και αποτελεί κοινή προσπάθεια της Γενικής διεύθυνση ένταξη και Ιστορικών Υποθέσεων της Ένωσης και βέβαια και του ΩΣΑ. Η ένταξη των μεταναστών και των παιδιών τους αποτελεί ε, μια πολύ μεγάλη ανησυχία για όλες τις χώρες του ΩΣΑ. Είναι καιροί που συνιστούν πολλές προκλήσεις και πολλά θα εξαρτηθούν εν μέρη και από τη μοίρα που επιφυλάσσουμε στους μετανάστες και στα παιδιά τους στις χώρες μας. Η χώρα αυτή παρουσιάζει λοιπόν τα πορίσματα ε, περί ένταξης των μεταναστών ε, και διασκεδάζει και κάποιους μύθους, κάποιες ε, ε, προκαταλήψεις για αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Οι μετανάστες είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας. Σχεδόν ένα στους πέντε κατοίκους των χωρών της Ένωσης και του ΟΣΑ είναι ή αλλοδαπός, έχει γεννηθεί δηλαδή σε άλλη χώρα, ή έχει γεννηθεί μεν στη χώρα αυτή που ζει, αλλά ένας από του δύο γονεί του αλλοδαπή. Πάνω από 30% αύξηση έχει σημειώσει ο αριθμό ε, των ε, μεταναστών το 2000 και μετά και αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπολείπονται ε, των ε, ατόμων που έχουν γονείς ε, γηγενείς. οι μεταναστές σε όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η παιδεία, εδώ συνοδεύομαι σήμερα από τον συνάδελφο Στέφανο Σκαρπέτα, που είναι ο Διευθυντής ε, της Διεύθυνσης ε, Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΩΣΑ και είναι και ο υπεύθυνος για αυτή τη δημοσίευση, για αυτό το έγγραφο. Ο Κριστόφ είναι ο συντάκτης του, που κάθεται εκεί κάτω. Μαζί με την ομάδα του βέβαια. Και μπορούν να απαντήσουν τα ερωτήματά σας στη συνέχεια, συνάδελφοι. Σχεδόν όλες οι χώρες ε, έχουν να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσεις ε, με τις νέες αφήξεις και χαμηλότερα αποτελέσματα σχεδόν παντού. Όπως επίσης ανάγκη προσαρμογής των μεταναστών στις χώρες υποδοχής Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, χώρες που γενικά θεωρούνται πολύ επιτυχημένες ε, ως προς την ένταξη των μεταναστών και εκεί βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την ένταξη αυτών των οφηχθέντων στις αγορές εργασίας είναι χαμηλότερα τα επίπεδα σε σχέση με τους ντόπιου. Και φαίνεται και από τα στοιχεία γιατί και πώς. Επίσης, οι μετανάστες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνήθως ε, ε, έχουν και λιγότερα ποσοστά απασχόλησης ό,τι αφορά ε, τους ντόπιου. Όσο πιο χαμηλά όμως είναι τα προσόντα τους, έχουν περισσότερες θέσεις αλλά κακής ποιότητας αυτοί που έχουν διπλώματα και προσόντα έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με τους ε, ντόπιου. Σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και αυτοί που έχουν ε, δεξιότητες και γλωσσομάθεια είναι άτομα με υπερβολικά υψηλά προσόντα για τη θέση που κατέχουν. Άρα θα μπορούσαν να κατέχουν κάποια καλύτερη θέση από αυτή που έχουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν διπλάσιοι είναι αυτοί. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών που σχετίζονται με, την, με το αντιστάθμιζα της απορρόφησης των μεταναστών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα επίπεδο εκπαίδευσης, κατηγορία, εργασία, οικογένεια. Είναι ανθρωπιστικός ο λόγος, είναι οικονομικός μετανάστης, ε, ήρθε γιατί ε, είναι εκτοπιστής κτλ. Και μπαίνουν σε διαφορετικά κουτάκια, σε διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχουν χώρες που έχουν περισσότερους ανθρωπιστικούς μετανάστες από ότι άλλους. Οι χώρες Σκανδιναβίας, για παράδειγμα, χρειάζονται αυτοί οι μετανάστες στήριξη και χρειάζεται και μια πολιτική ένταξη που μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να μην σας εκπλήσει. Βλέπουμε επίσης μετανάστες που είναι για μακρότερο χρονικό διάστημα στη χώρα να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και θα έλεγε κανείς ότι είναι λογικό αυτό, τώρα το τεκμηριώνουμε. Η πρόοδος δεν φαίνεται να είναι και σημαντική σε χώρες όπου οι πρόσφατες ε, ε, αφήξεις δείχνουν ότι εκεί υπάρχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Ολλανδία, Σουηδία, Γαλλία. Σε αυτές τις χώρες οι πληθυσμοί τα πάνε καλύτερα. Να περάσω τώρα σε κάποιες άλλες διαφορές. Για παράδειγμα, η οικονομική κατάσταση στη χώρα υποδοχής θα θεωρούσατε ότι είναι καθοριστικό παράγον. Ναι, θα μου πείτε, φυσικά. Και σίγουρα έχει και τον ισχυρότερο αντίκτυπο για τους μετανάστες. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να επηρεάζει τους ντόπιου. Ίσως γιατί είναι πιο κυκλική η φύση, αν θέλετε. Η Νότια Ευρώπη αντιμετωπίζει πιο μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ε, ένταξης των μεταναστών. Πολλοί έχασαν τις θέσεις του 10 της και όσοι εξακολουθούν να δουλεύουν, πάνω από το ίμιση δουλεύουν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, άρα αντιμετωπίζουν και ψηλό κίνδυνο φτώχειας, παρότι έχουν δουλειά. Δηλαδή μπορεί να δουλεύουν μεν, αλλά και η δουλειά τους και η αμοιβή τους κινδυνεύουν. Άρα θα είναι φτωχοί παρότι δουλεύουν. Και αυτό βέβαια σχετίζεται και με κακές συνθήκες ε, διαβίωσης, ε, στέγασης, ε, πολύ λίγα τα επιδόματα που παίρνουν κτλ. Έλλειψη ένταξη λοιπόν στην αγορά εργασία και κοινωνική ένταξη λυπής. Αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και τους ίδιους μετανάστες, αλλά και τα παιδιά τους. Πράγματι, το πιο ανησυχητικό πόρισμα του δημοσιεύματος αυτού είναι ότι και τα παιδιά που ε, γεννιούνται στη χώρα επηρεάζονται αρνητικά, παραδείγματος χάρη στον τομέα της εκπαίδευσης, από τις εισοδηματικές αυτές διαφορές. Δηλαδή, μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ε, η οικονομική αδυναμία, η κοινωνική αδυναμία από το γονέα στο παιδί. Αυτό το βλέπουμε στις ε, ευρωπαϊκές χώρες που οι μετανάστες είχαν λίγα προσόντα, λίγες δεξιότητες και πολλές φορές ε, μεταλαμπάδευσαν εντό αγωγικών την κοινωνία αυτή στα παιδιά τους. Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο ε, για να σπάσει η διαγενειακή μετάδοση αυτού του μειονεκτήματος. Όμως τα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά δεν έχουν τα μέσα ε, για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή. Στην ηλικία των 15 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Ισπανία. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, εκπαιδευτική επιδόσεις των ε, παιδιών μεταναστών που έχουν γεννηθεί όμως στη χώρα είναι χειρότερες από αυτές των ε, παιδιών που και οι δύο γονείς τους ε, είναι από την ίδια χώρα κατά ένα έτος. Δηλαδή σαν να έχουν φοιτήσει για ένα παραπάνω χρόνο από τις υπόλοιπες. Και τα παιδιά αυτά ουσιαστικά ε, δεν είναι ότι έφτασαν στη χώρα υποδοχής από τη Λατινική Αμερική, την Αφρική ή την Ασία. Έχουν πάει σχολείο, γεννήθηκαν και έχουν όλη τη ζωή και την έχουν ζήσει στη χώρα αυτή και παρόλα αυτά είναι ένα χρόνο πίσω από τα άλλα παιδιά λόγω αυτού του φαινομένου της μετάδοσης των μειονεκτημάτων και επειδή δεν σπάμε αυτό το φαύλο κύκλο. Άτομα τα οποία μεταναστεύουν ως ενήλικοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες επειδή μεγάλωσαν ε, ε, και σπούδασαν αλλού στις χώρες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Για τα παιδιά τους όμως δεν ισχύουν οι ίδιοι λόγοι. Γι' αυτό και αυτό το φαινόμενο τόσο λυπηρό. Και έχει να κάνει με, τη, τα εκπαιδευτικά συστήματα ε, που, και τις κοινωνίες των χώρων υποδοχής που θα πρέπει να φροντίσουν, να αφομοιώσουν τα παιδιά αυτά. Γιατί αλλιώς αυτό θα ήταν ηθικά, ε, η συνέχιση αυτής της κατάστασης ήταν και πολιτικά επικίνδυνη και ηθικά απαράδεκτη και κοινωνικά απαράδεκτη και είναι και ένα εμπόδιο προς την ανάπτυξη για όλους ε, κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή. Ενώ έτσι χάνονται και πολλές ευκαιρίες και στο μέτωπο της οικονομίας. Τα παιδιά των μεταναστών στην Ευρώπη έχουν σχεδόν, θα έλεγε κανείς, μόνο τις μισές ευκαιρίες να είναι πάνω στο 25% των ε, ε, καλύτερων μαθητών των σχολείων σε σχέση με τα παιδιά γονέων που μπορεί να προήλθαν από σχετικά μειονεκτικό υπόβαθρο, αλλά έχουν γεννηθεί στη χώρα και οι γονείς. Και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Ένα στους πέντε νέους με γονείς μετανάστες είναι νίτς. Δηλαδή δεν είναι ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην επαγγελματική κατάρτιση, ούτε ε, σε κάποια περίοδο, ούτε κάποια περίοδο μαθητείας. Και αν φτάσουμε μετά τα 15, ένα στους τρεις είναι η αναλογία η αντίστοιχη. Με αποτέλεσμα της ελλείψης αυτές, την ένταξη και τα προβλήματα ένταξης, υπάρχει μεγάλη αίσθηση διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των ατόμων ε, που ε, έχουν γεννηθεί από γονείς μετανάστες, αλλά στη χώρα υποδοχής Δηλαδή νιώθουν ότι υφίστανται διακρίσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάνω από ένα στους πέντε νιώθει ότι υφίστανται διακρίσεις. Είναι μεγαλύτερος δε αριθμός από αυτών που βλέπουν στου γονεί του, μετανάστες του ίδιου. Τα παιδιά νιώθουν ότι υφίστανται περισσότερε διακρίσεις από τους γονείς του. Αυτό είναι μια αποτυχία. Επίσης, αυτή η αίσθηση διακριτική μεταχείρισης είναι πιο έντονη σε αυτούς με καλύτερο μορφωτικό επίπεδο. Μπορεί να το καταλάβει κανεί γιατί ίσως ε, κανείς έχει περισσότερε προσδοκίε αφού έχει κάνει σπουδέ και μετά απογοητεύεται. Είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα αυτά. Και πρέπει να δράσουμε. Κυρίως οι χαράκτες ε, πολιτικής και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις, όπως εσείς οι πολιτικοί. Ίσως είναι, θα το πω να το πούμε μια στιγμή, Σπούτνικ. Ποτέ δεν ξέρει κανείς πάρα πολλά για αυτό το φαινόμενο, αλλά για πρώτη φορά ξέρει για αυτό το φαινόμενο χάρη σε αυτό το δημοσίευμα Πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που έγινε. Έχουμε πλέον την πρώτη ε, προσπάθεια να χαρτογραφήσουμε το τοπίο σε αυτό το τομέα που δεν είχαμε πολλές πληροφορίες. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, η χώρα υποδοχής ενός μετανάστη ή των παιδιών του. Επηρεάζει και τις ευκαιρίες που θα προσθέσουν στη ζωή. Όταν ο πρόεδρος Ομπάμα πρόσφατα είπε το μέλλον σας δεν μπορεί να εξαρτάται από το zip code, από τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Αυτό έχουμε εδώ όμως. Απλά δεν μιλάμε για ταχυδρομικό κώδικα, αλλά για τη χώρα καταγωγής πια Παρά τη σημαντική πρόοδο, σε πολλές χώρες πολλά απομένουν να γίνουν, Ιδίω για να έχουν οι μετανάστες και τα παιδιά τους τη δυνατότητα να πετύχουν στη ζωή, να βελτιώσουν την ένταξη, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουν ένα μέλλον ευημερία για όλους. Οι προκλήσει δεν είναι ανυπέρβλητε, αγαπητοί φίλοι. Οι Ευρωπαϊκέ χώρε και άλλες χώρες τόσα έχουν σημειώσει πρόοδο στην ένταξη. Περισσότεροι μετανάστες και τα παιδιά τους είναι καλύτερα ενταγμένοι στην αγορά εργασίας και στις κοινωνίες, χωρίς να σημαίνει όμως ότι είναι και καλά ενταγμένοι. Πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν. Η επιτυχής ένταξη σημαίνει καλύτερη δυνατή χρήση του δυναμικού των μεταναστών να αξιοποιηθεί το καλύτερο δυνατό που έχουν και να φτεθεί αυτό στην υπηρεσία τόσο των ιδιών όσο και της κοινωνίας στην οποία ζουν. Να συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια και να συνεχίσουμε να βλέπουμε τελικά πώς εντάσσονται οι μετανάστες στις χώρες μας. Settling in, εγκατάσταση, καλύτερα. Πότε έγινε το πρώτο, settling in το 2012, αυτό είναι το δεύτερο αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να είναι κοινή προσπάθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας. Ήταν προνόμιο για μένα το ότι ήρθα εδώ να σας παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία. Ελπίζω να ε, κατάφερα και να σας συναρπάσω αλλά και να σας ανησυχήσω ταυτόχρονα. Αλλά να ζητήσω και την υποστήριξή σας θα ήθελα για να συνεχιστεί αυτό το έργο και να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε κάτι που δεν θα φύγει ποτέ, αλλά μπορούμε πιστεύω να τα πάμε καλύτερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη Γενική Διεύθυνση Home, ε, η εκπρόσωπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται που δημοσιεύει την έκθεση αυτή σήμερα μαζί με τον ΩΣΑ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΩΣΑ που παρίσταται εδώ σήμερα για να παρουσιάσει την έκθεση. Όπως ξέρετε η μετανάστευση είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα και είδαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πόσο δύσκολες είναι οι συζητήσεις για κάποιες πτυχές για τη νέα ατζέντα για την μετανάστευση. Πάντα όμως τονίζουμε τις προτάσεις επανα εγκατάστασης τμήμα του πακέτου και βασικό τμήμα είναι η ενσωμάτωση των μεταναστών και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, όσους καλωσορίζουμε στην κοινωνία μας δεν θέλουν να μείνουν ως αποδέκτες βοήθειας. Θέλουν και αυτοί να συμβάλλουν σε αυτή την καινούργια ζωή μακριά από τον φόβο της δίωξης. Ε, και αυτό ισχύει για όλους τους μετανάστες, ανεξάρτητα των λόγων για τον οποίο ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η η ενσωμάτωσή τους λοιπόν θα καθορίσει και την επιτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά είναι και βασικός παράγοντας για την επιτυχία της Υπήρου μας. Ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη για την ενοποίηση, για την ενσωμάτωση των ε, μεταναστών στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο είχαμε το Ταμείο για την ε, ενσωμάτωση και στη νέα περίοδο για την ενσωμάτωση περιμένουμε να έχουμε 600 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά θέματα νόμιμης μετανάστευσης και ε, ενσωμάτωσης και το Κοινοβούλιο τονίζει πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο αυτό το 20% τουλάχιστον των ταμείων ε, για την άσυλο και τη μετανάστευση και την ε, ενσωμάτωση θα πρέπει να τα από τα μελη και αν δεν τα το ποσοστό αυτό θα πρέπει να το εξηγούν αυτό σε εσά και στους Ευρωπαίους πολίτες. Κάνουμε επίση ε, προσπάθειες την τελευταία δεκαετία να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικότερο ρόλο για την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ενσωμάτωση. Πριν από 10 χρόνια τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν κοινέ αρχέ για την ε, ενσωμάτωση και πριν από 5 χρόνια υπό την Ισπανική Προεδρία τα κράτη-μέλη συμφώνησαν επί κάποιων δικτών για να μετράται αυτή η προοδό για την ενσωμάτωση. Στη Σαραγώσα λοιπόν ληφθήκε αυτή η απόφαση και ως εκ τούτου είναι γνωστή ως δείκτες της Σαραγός. Αυτοί οι δείκτες λοιπόν ε, χρησιμοποιούνται σήμερα στην έκθεση. Η έκθεση είναι πάρα πολύ πλούσια σε υλικό και είμαι βέβαιη ότι θα χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο το 2014 για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι χώρες να καταρτήσουν μια πιο αποτελεσματική πολιτική για τους μετανάστες. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές και ο προλαλή σα τόνισε πολλέ εξ αυτών. Θα ήθελα εγώ να τονίσω κάποια ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, ε, το ποσοστό απασχόληση για τους υπηκός τρίτη χώρας είναι το μισό. Αυτό αφορά δύο τρίτα των μεταναστών και ένας στόχος της Ευρώπης ε, της 2020 αφορά ακριβώς την αποσχολησιμότητα. Βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020 ε, βάζοντας στο στόχο άστρο το θέμα της ε, απασχόλησης των μεταναστών. 18% έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης στις ηλικίε 25-34. Ε, Αυτό αντιστοιχεί σε επίπεδο δημοτικού και 4% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στους υπηκόους της χώρας, αλλά όπως ακούσαμε η καλή εκπαίδευση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα δαμειφθεί η καλή εκπαίδευση, δηλαδή στην αγορά εργασίας 64% των υπηκών τρίων, τρίτων χωρών με ε, ψυχείο πανεπιστημίου είχαν ε, δουλειά αντίστοιχη των ικανοτήτων Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των υπηκών της χώρας είναι 83%. Και ύστερα έχουμε και μεγάλη διαφορά για όσους έχουν πάρει το πτυχίο τους εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις συζητήσεις που γίνονται για τους ερευνητέ και για τους φοιτητέ και τη σχετική οδηγία. Αυτό σημαίνει μεγάλη απώλεια ικανοτήτων και για τα άτομα αλλά και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η κακή κατάσταση στην αγορά εργασία έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Το 2013 το ίμιση περίπου των υπηκών τρίτων χωρών ήταν σε κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού. Διπλό το ποσοστό αυτό σε σχέση με τους υπηκόους της χώρας. Εξηγείται επίσης ε, στην έκθεση ο βαθμός τον οποίο αντιλαμβάνονται ε, ή θεωρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών ότι υπόκεινται διακριτική μεταχείριση. Τα απορίσματα και τα ευρήματα είναι πολύ άριθμα και πολλά εξ αυτών ε, μας δίνουν όμως και ε, μια ελπίδα. Για παράδειγμα, οι προκλήσεις για την ενσωμάτωση δεν αυξάνονται με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών. Οι χώρες που έχουν ε, μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην ενσωμάτωση. Το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι τονίζεται. Επίσης, μπορούμε να μάθουμε το εξή από την έκθεση, ότι η ενσωμάτωση είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία, αλλά με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα χάσματα και τα μειονεκτήματα. Είναι πολύ πιο προφανή για πρόσφατους μετανάστες, ενώ όσοι οι μετανάστες είναι στην Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια έχουν πολύ πιο καλά αποτελέσματα να επιδείξουν και πιο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πιο πολλοί μετανάστες είναι ενεργοί πολίτες. Το 2013, δύο τρίτα των όσων είχαν γεννηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν λάβει την υπηκότητα μετά από 10 χρόνια παραμονή στη χώρα και 10... 70% ψήφισαν στις τοπικές εκλογές. 70% για πολλές χώρες αυτό, για χώρες που δεν είναι υποχρεωτική η προσόλευση της κάλπος είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα για τα κράτη-μέλη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σημειώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά για την ενσωμάτωση, θέλουμε να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συζητήσεις μας. Χαίρομαι που υπάρχει πλέον μια σταθερή και καλή βάση δεδομένων, βάση της οποίας θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε και πάλι τον ΩΣΑ για την καλή δουλειά που κάνουν για την ενσωμάτωση και για την νόμιμη μετανάστευση, όπου συζητάμε προσφάτως ε, το θέμα ότι όλα αυτά τα συζητάμε και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον ΩΣΑ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, αλλά έχω τρει συναδέλφου που θέλουν το λόγο. Του τον δίνω. Αναγκόμεση στην πρώτη. Ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση και την έκθεση. Είναι συναρπαστικά τα δεδομένα που περιλαμβάνει. Το μόνο που ελπίζω είναι να φροντίσετε να τη δουν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διότι το χρειάζονται αυτό. Το λέω, διότι η τελευταία συζήτηση στο Συμβούλιο ήταν τελείως παράλογη, ήταν απαράδεκτη. Και δεν αφορούσε την Ελλάδα, αφορούσε τη μετανάστευση. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη μετανάστευση ζητήθηκαν. Οι ε, κύριοι λοιπόν αυτοί και οι κυρίες αυτές πρέπει να καταπιούν από το βιβλίο. Πρέπει κάποιο να το χώσει στο λαιμό. Και καλό θα ήταν να σα ακούσαν, να σας ακούγανε. Μπα και καταλάβουν ότι ο μόνο τρόπο να σταματήσουν οι τραγικέ καταστάσει που γνωρίζουμε στη Μεσόγειο αλλά και σε άλλα μα σύνορα, ε, χερσαία, ο μόνο τρόπο να δώσουμε τέλος στην λαθρεμπορία και τα δίκτυά τη είναι να προβλεφθούν νομίμες οδοί για την μετανάστευση. Επίσης πρέπει να επισημάνω ότι οι διστακτικές αντιδράσεις πολλών από, τον, από τις κυβερνήσεις μας έχουν να κάνουν και με την διάθεση που επικρατεί στις κοινωνίες μας οι οποίες έχουν αρχίσει να φοβούνται. Φοβούνται τους μετανάστες. Παρόλο που όπως δείχνει το βιβλίο σας, τους χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Τους χρειαζόμαστε για μια σειρά από λόγους, κυρίως για την αποτελεσματικότητά μας στην οικονομία και είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή στην Ευρώπη και για την πρόοδο. Ακόμη και για την εξισορρόπηση των λογαριασμών της κοινωνικής ασφάλειας, της κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό ίσχυε στη χώρα μου οπωσδήποτε έω το 2008. Απλώ το 2008 με την κρίση Το επίπεδο των μεταναστών στην Πορτογαλία μειώθηκε δραματικά κατά 10 φορές και αυτό που αυξήθηκε ήταν η μετανάστευση από την Πορτογαλία εξαιτίας της παράλογης και χωρίς λογικής της τυφλής λιτότητας που επιβλήθηκε από την Τρόικα και που επέλεξε η κυβέρνησή μας. Τώρα τι έχουμε. Ελπίζω ότι η επόμενη σας έκθεση και σας το ζητώ αυτό κυρία, κύριε Γκουρία και σας εσάς κυρία Πάικ από την Επιτροπή να καταγραφούν στοιχεία για τις συνέπειες της πολιτικής λιτότητας ως προς την μετανάστευση από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και την διαρροή γεφάλων. Διότι αυτοί που έχουν φύγει είναι κυρίως ανθρώποι με πολλά προσόντα, με υψηλά προσόντα, νέοι που τους χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη. Στην περίπτωση μιας χώρας όπως η Πορτογαλία πρέπει κανείς να πάει μια πεντηκονταετία πίσω για να δει το ίδιο επίπεδο μετανάστευση από τη χώρα ε, που βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια. Πάνω από 3.000 Πορτογάλοι έφυγαν για να μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Και η άλλη μου ερώτηση είναι ότι σημειώνω αυτά που λέτε κύριε Γενική Γραμματέα, τα σημαντικά πορίσματα για την ε, αίσθηση του να είναι κανείς αποκλεισμένος, ιδίως μεταξύ των παιδιών των μεταναστών φαίνεται να είναι ένα ποσοστό 1 έως 5%. Είναι πολλοί κόσμος αυτό. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι, όλα τα μέλη ε, εντελώ, είναι ότι οι πολιτικές τους προκαλούν τον κοινωνικό αποκλεισμό με τις πολιτικές λιτότητας, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά όχι μόνον. Και τελικά αυτό που παράγουμε είναι ότι παράγουμε ξένους μαχητές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να περιοριστείτε όμω τα δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σα, διότι μα τελειώνει ο χρόνο. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Η κυρία Σίπελ. Παρακαλώ, all, Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά για όλες αυτές τις εκθέσεις και όλα αυτά τα δεδομένα για τα πιο πολλά από αυτά που ακούσαμε εδώ στη συνάντηση δεν είναι καινούργια, αλλά στην πολιτική συζήτηση μας λείπουν σε κάποιες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα δεδομένα, τα στοιχεία για να αποδείξουμε την ε, κατάσταση. Και είναι λυπηρό το να αναφέρουμε ότι στα κράτη-μέλη μας, αν ε, οι γονεί σου είναι φτωχοί, είσαι και εσύ φτωχό. Αν οι γονεί σου είναι ανειδίκευτοι, θα είσαι και εσύ ανειδίκευτο. Και έτσι παρατείνονται οι καταστάσει. Τέτοιε, Είναι λυπηρό λοιπόν πραγματικά αυτό στα κράτη-μέλη και είναι λυπηρό που τα κράτη-μέλη δεν εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και αληθεύει επίσης ότι αυτό είναι πολύ χειρότερο για τα παιδιά των μεταναστών. Συμφωνώ. Είναι απαράδεκτο αυτό σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο στοιχείο, την οικονομική κατάσταση και, πιστεύω ότι αν μιλάμε για τα παιδιά των μεταναστών, αυτή η κατάσταση διαρκούς ευθυντικής μεταχείρισης σε όλους τους τομείς έχει και επιπτώσεις για ένα φαινόμενο που μας απασχολεί πολύ, την ρίζοσπαστικοποίηση, γιατί προφανώς αισθάνονται πιο πολύ ότι ε, δέχονται διακριτική μεταχείριση τα παιδιά αυτά είναι γεννημένα εδώ πέρα και πιστεύουν ότι είναι τμήμα και πολίτες της χώρας αυτής. Και ύστερα επανελειμμένα ε, διαπιστώνουν ότι αυτό δεν στέκει. Άρα, είναι πολύ και πολυεπίπεδοι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Χαίρομαι που έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας πλέον και ελπίζω αυτό να έχει κάποια κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τους μετανάστες, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δουλέψουμε και για τα δικά μας παιδιά, για τους δικούς μας πολίτες. Αλλά συμφωνώ, όταν πρόκειται για τους μετανάστες, τα παιδιά μεταναστών, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δεινή και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη που συμπλέει με τις ακροάσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα όπου ο κύριος Μάρτιν και ο κύριος Βυσέλτη πρόσθε... επεσήμαναν την προστιθέμενη οικονομική αξία της νόμιμης μετανάστευσης και το γεγονός ότι στις χώρες όπου υπάρχει πραγματική εργασία και ε, η σωστή ένταξη των μεταναστών αυτό ωφελεί τους πάντες. Είναι σαφές από τη μελέτη σας και το είπατε πολύ ξεκάθαρα και την ε, προηγούμενη φορά και πάντοτε μας εκπλήσουν αυτές οι δύο διαφορετικές εκδοχές ως προς το φαινόμενο της μετανάστευσης, δηλαδή ο έλεγχος των συνόρων και το οικονομικό του άκτος ή εάν πρέπει η πρώτη προτεραιότητα να είναι η νόμιμη η μεταναστευση και η κοινωνική ένταξη μαζί με τα οικονομικά της ωφέλη. Ελπίζω, όπως είπαν προηγουμένως η Άννα και η κυρία Σίπελ, ότι η μελέτη αυτή θα αναγνωστεί ε, επανειλημμένως διότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και από οικονομική σκοπιά έχει ενδιαφέρον για όλου για όλους του Ευρωπαίου πολίτε, ε, για αυτού που έφτασαν ε, πρόσφατα ή αυτού που είναι εδώ από καιρό. Δεν έχει σημασία αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η κυρία Λάβριστην. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Όσα για αυτό το βιβλίο. Διότι Έχω ασχοληθεί με τα θέματα της μετανάστευσης και τη σχετική έρευνα από το 1997 και την περιμέναμε, τη λαχταρούσαμε αυτή τη μεγάλη συγκριτική μελέτη με την εικόνα που παρουσιάζει. Αυτό που μου λείπει όμως εδώ, ίσως, είναι μια συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών ένταξη στις διάφορες χώρες. Διότι αν δούμε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες, είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε εάν δούμε τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών ένταξη. Ο έχει κάνει πολύ συγκριτική δουλειά ε, από πολιτική οπτική γωνία. Εδώ θα ήταν μια καλή ιδέα για τη, για τη μελλοντική σας έρευνα να δείτε τις πολιτικές ένταξεις ή το κατά πόσον αυτές δεν υπάρχουν. Και παράλληλα, σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η το κατα ποσον αυτέ δεν υπαρχουν και παραλληλα σημαντικο ειναι κατάσταση ως προς την οικονομική διάσταση Ίσως λείπει ο δείκτης της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ίσως να μπορούσε να υπάρχει και ένας δείκτης ένταξης, γιατί οι δύο προσεγγίσεις που ακολουθούνται εδώ ίσως να μην αρκούν. Ίσως πρέπει μόνοι μας να καταρτήσουμε ένα τέτοιο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης και να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τις διάφορες πολιτικές μας προτεραιότητες. Ε, και εδώ θα ήταν ίσω ένας καλό τρόπο αυτό να αντιμετωπίσουμε όλων των ειδών τα στερεότυπα. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια συγκριτική εικόνα με τους συγκριτικούς πίνακε. ευχαριστούμε. Η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ τους συντάκτες και τους ε, ομιλητές μας για την ε, παρουσίαση τη μελέτης αυτής. Εγώ, υπουργό μετανάστευση. Θα ήθελα να έχω μαζί μου ένα παρόμοιο έγγραφο για να αποδείξω ότι έχω κάνει τόσα χρόνια και χαίρομαι που σήμερα βλέπω ότι αυτό το βιβλίο ε, δημοσιεύεται και μπορείτε να μας το παρουσιάζετε. Αυτό το κείμενο μα φέρνει αντιμέτωπο με το γεγονό ότι υπάρχει ένα γεγονό που πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίσουμε τι πολιτικέ μα τι κατεπίγουσε ανάγκε. Όταν τα αναλύουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι το φαινόμενο τη μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο διαφορετικό. Τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ε, απαραίτητο να βρούμε συγκεκριμένου πόρους για να τα αντιμετωπίσουμε. Και επίσης σκόπιμο και απαραίτητο είναι να έχουμε μια κοινή θεώρηση και των πολιτικών για την ένταξη που να μετατραπεί ε, σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένε δεσμεύσει. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω βάση για να εκμεταλλευτούμε όλες τις καλές πρακτικές για την κοινωνία των πολιτών, θεσμικά όργανα, ε, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αξιοποιούνται επαρκώ, διότι ξεκινώντα από αυτήν την ε, αφετηρία θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα προγράμματα και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, οργανικής αξίας που να έχει περισσότερο νόημα και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Οι ίδιες οι πολιτικές της μετανάστευσης πρέπει να ενταχθούν στην κοινότητά μας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια ευκαιρία για να σκεφτούμε από κοινού πώς οι πολιτικές μετανάστευσης μακροπρόθεσμα με ε, ελεγμένα στοιχεία όπως αυτά που μας παρουσιάζεται σήμερα μπορούν να εμπνέονται από μια ευρεία και οργανική θεώρηση του τι συμβαίνει στην πράξη, στις περιφέρειες και τις κοινότητες. Δηλαδή από την εθνική πραγματικότητα του κάθε ώστε να σχηματιστεί ένας κοινό ευρωπαϊκός και διεθνής ορίζοντας. Αυτός είναι ο στόχος. Χαίρομαι που άκουσα τις προαλήσεις σας συναδέλφους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να αξιοποιήσουν αυτή τη μελέτη και να σχεδιάσουν πολιτικές μετανάστευσης, οι οποίες να μας οδηγήσουν σε καλύτερη συνύπαρξη των κοινοτήτων που συνεπάρχουν στις διάφορες επικράτειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κουρία, θέλετε να απαντήσετε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ Μπελίντα και σένα για την παρουσίασή σου. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική και δείχνει εκτός μικροφώνου ο ομιλητής. Απλώς όλα αυτά προχωρούν σταδιακά γεωμετρικά. Ε, παράγουμε μαζί πολύ καλή δουλειά, ε, καλά αποτελέσματα και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες είπε ότι θα πρέπει να κοπανίσουμε τα κεφάλια των μελών του Συμβουλίου ε, με, αυτό το βιβλίο. Ε, τους δίνουμε αντίγραφα, ακολουθούμε πιο φιλινικές μεθόδους. Και θα φροντίσουμε και οι συνεργάτες τους να λάβουν αντίγραφα και κλίδες USB για να τα δουν και στις οθόνες τους αλλά θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν οι ηγέτες. Αυτούς θα τα στείλω στους ε, αρχηγούς κυβερνήσεων του G20, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, σε όλους τους υπουργούς και σε όλους τους σχεδιαστές πολιτικές τους υπουργούς, τους γενικούς διευθυντές, πρέπει αυτοί να εκθέσουν τις πολιτικές επιλογές στους επικεφαλείς. Θα το προωθήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καταλάβετε νομίζω το εξή. Όλοι ε, δεν ξέρουν πώς να βρουν λύση. Όλοι αισθάνονται δυσάρεστα και ε, ε, μένουν άναυδοι λόγω του όγκου των διαστάσεων, της ισχύω, της δύναμης κρούσης και των αριθμών που καταγράφουμε δεν εκπλήσωμε από στο του Συμβουλίου, τελείωσε με τόνους έντονους, διότι το ερώτημα εδώ δεν είναι απλώς αν έχουμε μια καλή πολιτική μετανάστευση ή όχι. Έχει να κάνει με τα θεσμικά όργανα, έχει να κάνει με την ετοιμότητα, έχει να κάνει με το αν η Λιβύη καταραίει η Συρία, καταραίει εάν εκατομμύρια άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα, τι κάνουμε. Αυτή δεν είναι μετανάστευση που θέλει, ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν εδώ. Ούτε είναι άνθρωποι που ειρηνικά θα εγκατασταθούν και θα κοιτάξουν να πάνε σχολείο και πανεπιστήμια τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι αυτοί απλώς φοβούνται για τη ζωή τους, σε καθημερινή βάση. Οπότε λίγο διαφορετικά το φαινόμενο είναι ελαφρώς διαφορετικό. Ναι, ε, πρέπει να πω ότι μέχρι αυτές τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες και μήνες οι λογαριασμοί μας ήταν πολύ σαφείς. Καθαρός φορολογικός αντίκτυπος. Αυτό σημαίνει στις κοινωνίες μας η μετανάστευση είναι εποφελής. Δεν κοστίζει στους φορολογουμένους. Και είχαμε τεκμηριώσει αυτό το στοιχείο και η Σεσίλια Μάρθον και ο Λάσλο Άντορ πριν από δύο χρόνια ήδη είχαν παρουσιάσει την πρώτη αριθμητικών δεδομένων, λέγοντας ότι αυτό είναι το καθαρό φορολογικό κέρδος. Αυτό που συμβαίνει επίσης είναι ότι όταν έχει κανείς περισσότερη ανεργία και μετά αυτή τη μαζική έλευση μεταναστών, Αυτά φυσικά και επηρεάζουν τα φορολογικά. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπήρχε εξισορρόπηση, να έγειρε προς την αμυντική πλευρά η ζυγαριά, αλλά σε γενικές γραμμές η μετανάστευση έχει αποδειχθεί επωφελής από φορολογική σκοπιά. Και σε πολλές περιπτώσεις με τη γύρανση του πληθυσμού η μετανάστευση είναι ο μόνος τρόπος για να τονωθούν και να συνεχίσουν να πτήσονται οι οικονομίες. Ε, η παραγωγικότητα θα συνεχίσει να, ε, μειώνεται, να ε, βελτιώνεται. Και δεν θα έχουμε καμιά άλλη επιλογή στο μέλλον αν δεν υπάρχει μετανάστευση γιατί η κοινωνία θα συρρυκνώνεται και οι πολιτικέ μετανάστευση μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο εύρωστη κοινωνία. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο καλή ποιότητα έχει η πολιτική ενταξή μα, όπω είπατε, Αναγκόμε. Τώρα, δεύτερο γιατί βλέπω τον συνάδελφο που μου λέει ότι πρέπει να βιαστώ, ένα στους πέντε είναι πολύ και ένα στους τρεις είναι ακόμα πιο πολύ. Είναι δύσκολο να πούμε ότι η σχέση θα γίνει ένας προς ένα, αλλά είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη λιτότητα. Δεν το πιστεύω αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η λιτότητα δυσκολεύει πολύ τα πράγματα, διότι απορροφά καταργεί, καταργεί κάποια τα κονδύλια, αλλά πρέπει να σχεδιάζουμε καλύτερα και τον προπολογισμό. Κυρία Ζήπελ, γεγονότα, ξανά γεγονότα και πάλι ε, γεγονότα. Ναι, ε, η προσέγγιση μας είναι κάπως ε, διαισθητική και με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις, όμως τα δεδομένα βοηθούν, επιτρέπουν να αποφύγουμε τις προκαταλήψεις στις συζητήσεις μας ή να υπάρχει ιδεολογική φόρτιση διότι ακόμη και με την κλιματική αλλαγή υπάρχουν άνθρωποι που την αρνούνται. Ε, οπότε θα πει κανείς πώς η επιστήμη να το αποδείξει. Η επιστήμη προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία καθημερινά. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζουμε ότι ξέρουμε, τελικά δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Με πιο οργανωμένο τρόπο για να έχουμε αποτελεσματικότερη μελέτη του θέματος. Η Άννα Γκόμες είπε ότι τα κράτη αποφασίζουν. Ναι, αλλά το σώμα αυτό ε, αποφασίζει επίσης και στέλνει τα ανάλογα μηνύματα στις διάφορες χώρες. Αυτοί αποφασίζουν τι θα κάνουν και τους δίνει μια πολιτική κατεύθυνση για να προχωρήσουν. Κυρία Νταλόν Μπονφά ή κάτι τέτοιο. Νταλόν Μπονφά, σωστά. Ωραία. Η μετανάστευση είναι αποφελής για όλους. Το ερώτημα είναι εάν θα υπάρχει έλεγχος ή αν αυτό το ε, αντιπαραθέτουμε ή μάλλον αν θα υπάρχουν επενδύσεις στα σύνορα και αυτό το αντιπαραθέτουμε με τις επενδύσεις για την ένταξη. Όπως το πρώτο είναι κάπως περιττό, διότι τελικά οι μετανάστες θα βρουν τρόπο να δυσδύσουν Σας το λέω ε, γνωρίζοντας πολύ καλά το φαινόμενο της μετανάστευσης διότι στη χώρα μου υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες που έφταναν, μάλλον ξεκινούσαν για να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένε Πολιτείε και στις Ηνωμένε Πολιτείε έχει πιο πολλούς Ισπανόφωνους από ότι νεύρους, ε, μαύρους Αφρικανούς και 12% του πληθυσμού είναι 36 εκατομμύρια. Είναι Ισπανόφωνοι, ισπανική καταγωγής, και ε, από αυτούς το 70% είναι ε, Μεξικάνοι, 25 εκατομμύρια Μεξικάνοι στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνω λοιπόν το θέμα, αλλά δείτε τι γίνεται. Ο τελευταίες μέρες ο Ντόναλτ Τραμπ αναφέρθηκε στη μετανάστευση και βλέπουμε να υπάρχει ε, μια αίσθηση ότι δεχόμαστε εισβολή. Μια αίσθηση ότι θα χάσουμε τα κεκτημένα μας. Δεν είναι όμως ο φόβος του να μοιραστεί κανείς. Είναι ο φόβος του να μοιραστεί το ίδιο, το ίδιο κομμάτι από το κέικ, από την τούρτα. Ε, το θέμα είναι ότι αν κόψουμε την τούρτα σε πιο πολλά κομμάτια η φέτα θα γίνει πιο λεπτή. Δεν είναι όμως έτσι το ερώτημα είναι πώς να εντάξουμε τους μετανάστες ώστε να ε, αναπτυχθεί η οικονομία, να πάρει άλλες διαστάσεις, να γίνει πιο ισχυρή, να πάρει ελβαρύτητα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι γι' αυτό θέτουμε το θέμα των προσόντων. Δεξιότητες, δεξιότητες, δεξιότητες, προσόντα, προσόντα, προσόντα. Αναβάθμιση των προσόντων. Άνα αναβάθμιση. Δεν μιλάμε μόνο για εκπαίδευση η εκπαίδευση, η, κατάρτι, η μάθηση, η κατάρτιση, η επαγγελματική κατάρτιση, ε, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν σχολεία και πανεπιστήμια αν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμός μεταξύ της δράσης των θεσμικών οργάνων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργαζομένων και των εταιριών αλλά και των κυβερνήσεων. Τελειώνει ο χρόνο μου, κυρία Λόρεστιν. Το θέμα των πολιτικών ένταξης. Συμφωνώ, η πολυδιάστατη προσέγγιση, αναγκαία κι αυτή, και ο δείκτης ένταξης. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε βαθμολόγηση και ιεράρχηση. Κυρία Κέγγε, να σας πω απλώς ότι συμφωνώ απολύτως. Το ζήτημα είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει πρώτα να γνωρίζουν για να συζητούν μετά, αλλά εν τέλει πρέπει και να αποφασίσουν κάποια στιγμή. Είναι σαφές αυτό. Εμείς πρέπει να θέσουμε επιτάπητος, εμείς όλοι μαζί, ε, το θέμα, γιατί τελικά οι ηγέτες και μόλις ξεκινούμε, τώρα είναι η αρχή. Γι' αυτό μπορεί και να έχουμε συζητήσεις λίγο πιο έντονες και να μην οδηγούμαστε σε οριστικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε που πρέπει να διακόψω την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση, αλλά είμαστε τελείως εκτός χρονοδιαγράμματος και έχουμε και άλλα σημαντικά σημεία στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας εδώ, να σας ευχαριστήσω για την εκθέση, για το έργο σας εν Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Παρουσία τη ετήσια έκθεση 2014. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Τζοβάνι Μπουταρέλη, ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία Δεδομένων, για να μα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση το 2014. Πρόκειται βέβαια για ένα έτος μετάβασης μεταξύ ε, τη νέα ομάδα που διορίστηκε, τη και τη νέας που διορίστηκε το Δεκέμβριο. Θέλω να ευχαριστήσω ε, για την ε, Ευχαριστώ σας καλοσύνη να είστε εδώ κύριε Μπουταρέλη και να σα συγχαρώ για το έργο που έχετε ήδη επιτελέσει εσεί και η ομάδα σα Θα σας δώσω το λόγο να μα παρουσιάσετε καταρχά την έκθεσή σα και έπειτα να ξεκινήσει η συζήτηση. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Σήμερα λίγη μια μεταβατική περίοδος για το θεσμό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ξανά σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω αυτή τη φορά την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου πόπτη Προστασίας Δομένου για το 2014. Σήμερα από τη συνέχεια περνάμε σε μια πιο ορατική θα έλεγα προσέγγιση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις για την ψηφιακή Ευρώπη. Η ευκαιρία του ορισμού μου, τον ε, συνάδελφό μου, τον αναπληρωτή, ε, τον ε, κύριο και εμένα, μας είπατε ότι πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να προτείνουμε συστάσεις και πρακτικές λύσεις. Ο Βότσεχ και εγώ Έχουμε πρακτική εμπειρία και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε ανεξάρτητες από ποιες αρχές. Θα θέλαμε λοιπόν να σας καλήσουμε, καλέσουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εμπειρία για να βρούμε λύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάμε μια φωνή για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να οικοδομήσουμε γέφυρες και με τους επανατλαντικούς μας εταίρους. Είμαι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσω και για κάποια πιο λεπτά ζητήματα όπως είναι τα Μητρώα Επιβατών, PNR, για τα οποία πλέον έχετε δώσει... Ε, έχει αναλάβει και δεν στο Συμβούλιο το συζητήσει, έχουν κατατεθεί εκατοντάδε από τροπολογίε, Είναι Ηράκλειο το έργο που αναμένει το εισηγητή Κέρκοπ για να καταλήξει σε μια συνεντική λύση. Όμως, αυτό που βασικά εμάς μας ανησυχεί στο επίπεδο του Ευρωπαίου Επόπτη είναι το γεγονός ότι από τότε που μας καλέσετε για τελευταία φορά να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το Γενάρη συγκεκριμένα, έχουν προκύψει στοιχεία. Μάλλον τα διαθέσιμα στοιχεία που να δείχνουν ότι χρειάζεται δημοκρατική ε, εποπτεία, δημοκρατικός έλεγχος, είναι πλέον διαθέσιμα σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων PNR. Εσείς είστε όμως οι νομοθέτες. Και άλλωστε η πολιτική είναι ε, η τέχνη του εφικτού. Εμείς θέλουμε να σας δώσουμε ειλικρινείς αμερόληπτες απόψεις σε σχέση με τις ενίοτε σοβαρές ε, επιπλοκές που μπορεί να έχουν ε, τα συλλογή αυτών των στοιχείων για την προσωπική ζωή των η προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια καλή ε, ιστορία. Το 2014, τα επόμενα χρόνια, θα το θυμάται κανείς ε, ως ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό έτος, γιατί η ιδιωτική σφαίρα, η προστασία δεδομένων από την νομική θεωρία πραγματικά πέρασαν στην πραγματικότητα. Για τη δική μας οργάνωση το 2014 ήταν ένα μεταβατικό έτος που χαρακτηριζόταν από αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την εκλογή και τον ορισμό ε, και τη θητεία μας. Από την έκθεση τώρα, η οποία διατέθηκε στη γραμματεία σας και τώρα νομίζω μπορείτε να τη βρείτε και ε, στην αίθουσα σε δύο διαφορετικές γλώσσες, διατηρήσαμε ε, τα επίπεδα των επιδόσεών μας Σημαντικές επίσης ε, αποφάσεις του δικαστηρίου είχαμε για την επιτήρηση και ιδίω για την ε, διακράτηση δεδομένων και την ε, σωστή, το σωστό χειρισμό και επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς λόγους. Έχουμε την Ισπανία Google κατά Ισπανία, το δικαίωμα στη λύθη όπως αποκαλείται και ούτω καθεξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης στήριξε τον αφαιρημένο κείμενο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, χαίρεται πολύ που μπορεί να βοηθήσει τους εισηγητές, τους και όντες εισηγητές στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Αν αναλύσουμε όμως τι έγινε πέρυσι, μπορούμε να πούμε ότι εσείς ε, που χαράσετε την πολιτική θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι κανόνες περί ε, ροής ε, δεδομένων μεταξύ Ευρωπαίων ε, και άλλων εταίρων. Και αυτό και πέρυσι τον Ιουνίο δημοσιοποιήσαμε μία γνωμοδότηση στην οποία Καλούμε το Συμβούλιο να διδαχθεί τα μαθήματα του παρελθόντος, να λάβει υπόψη του ε, τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, ε, αναπτύσσουμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν καλύτερα να εφαρμοστούν και να ενταχθούν στις πολιτικές ε, οι πολιτικέ υπερπροστασία δεδομένων. Καλούμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχθεί αυτή την ε, προσφορά. Πριν από τέσσερι μήνε δημοσιοποιήσαμε, όπω γνωρίζετε, τη στρατηγική για τη συνέχεια και την αλλαγή. Είναι ένα σταθερό σχέδιο και πρόγραμμα. Βασίζεται και στην εμπειρία του Βόιτσα και στη δική μου εμπειρία ω εθνικών εποπτών. Και βέβαια συνεργαστήκαμε στενά με τους εταίρου μα διμερό σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 των εξάρτων Αρχών Προστασίας Δεδομένων. Κυρίως ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χειρίζονται τις ε, υπηρεσίε προσωπικού χαρακτήρα, για το προσωπικό, για τους παραγωγούς κτλ. κτλ. Το 2014 ε, στον οργανισμό μας 144 γνωμοδοτήσεις δημοσιοποιήσαμε όπου ελέγχουμε διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. Είχαμε 210 καταγγελίες που αφορούσαν ορισμένες σημαντικά ζητήματα και κάναμε οκτώ επιτόπιες επισκέψεις, επιθεωρήσεις και σε Συμβούλιο Κομισιών Κοινοβούλιο εστιάζοντας ε, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ε, για να δημιουργηθεί μια νοοτροπία προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Στο Συμβούλιο, για παράδειγμα, εργαστήκαμε με το προσωπικό που παρέχει καθοδήγηση για, για θέματα όπως είναι η ε, μεταφορά δεδομένων και για ευαίσθητα θέματα όπως είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχει και ένα εργαστήριο πληροφορική το οποίο δημιουργήθηκε πέρυσι για να αξιολογεί το πώς επηρεάζουν την ιδιωτικότητα οι νέες τεχνολογίες και αν υπάρχει συμμόρφωση των ιστοσελίδων με του κανόνε περιπροστασία δεδομένων στου φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι ξεκινήσαμε να έχουμε έναν συμβουλευτικό ρόλο, ε, προληπτικό, ενεργητικό. Είχαμε και 46 άτυπα ή ε, επίσημα σχόλια. Δημοσιεύσαμε επίση και κάποια σημαντικά προκαταρκτικά έγγραφα, όπως για παράδειγμα πώς σχετίζεται ανταγωνισμός, ε, ο νόμος περί ανταγωνισμού και καταναλωτών. Έχουμε ε, μία εργαλειοθήκη επίσης και έχουμε συνεισφέρει και στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σε ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τα θεμητά συμφέροντα, οι νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την επιτήρηση κτλ. Επίσης, Έχουμε και μια πρωτοβουλία για ένα μηχανικής δικτύων μεταξύ ακαδημαϊκών, των πολιτών, ερευνητών, ακαδημαϊκών για να έχουμε πρακτικές μηχανικής engineering που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες μας περί προστασίας δεδομένων και θέλουμε και στις εφαρμογές και στις υπηρεσίες και στα προγράμματα οι προγραμματιστές να εισαγάγουν ε, παραμέτρους σχετικές με αυτή την προστασία δεδομένων. Να σας πω κάποια πράγματα για την προστασία δεδομένων. Εξακολουθούν να είναι τεράστιες οι προσδοκίες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη στους επόμενους μήνες. Εχθές 109 χώρες είδαμε ότι έχουν νόμους για την ε, ιδιωτικότητα. Στη μειοψηφία για πρώτη φορά οι ευρωπαϊκές χώρες. Τεράστια ευκαιρία. Πρέπει να αγηθούμε για τις πολιτικές αυτές ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων. Από την Ιαπωνία μέχρι τη Βραζιλία, από την Ινδία μέχρι την Αφρικανική Ένωση διάζονται νέα νομοσχέδια, καταρτίζονται νέα νομοσχέδια και τα είναι στραμμένα σε εμά. Ε, με προσέγγισαν αντιπροσωπείς από τη Σιγκαπούρη, το Μαρόκο, ε, τις Βερμούδες για να συζητήσουν τα σχέδιά τους μαζί μας να δουν τι αποφάσεις ε, μπορούμε εμείς να λάβουμε εδώ και να μας ακολουθήσουν, να μας μιμηθούν. Έχουμε τριμερή διάλογο τώρα για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Σωστή διαδικασία, αλλά όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι θα συνεπάγεται αυτός ο νέος νόμος. Δεν υπάρχει περιθώριο για σφάλματα. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση για την επόμενη γενιά πολιτών. Post-millennials ή η γενια Z. Είναι οι έφηβοι, τα παιδιά που γεννήθηκαν την τελευταία 15 ετία, που έχουν ζήσει ε, τη γενιά του διαδικτύου των οφωνών αφής από την ώρα που γεννήθηκαν. Και οι ίδιοι θα προγραμματίζουν την τεχνολογία, δεν τη χρησιμοποιούν μόνο, άρα πρέπει η μεταρρύθμιση να πετύχει και θα κρατήσει για τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να βάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στο κέντρο βαρύτητας. Αργότερα αυτό το μήνα λοιπόν ε, θα σας δείξουμε στην πράξη ότι είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε. Θα έχουμε ένα position paper ως ε, εφαρμογή ε, που θα μπορείτε να κατεβάσετε στα smartphone και στα κινητά και στις ταμπλέτες σας και θα είναι χρήσιμο για όλου όσου ενδιαφέρονται για αυτή την μεταρρύθμιση και όχι μόνο τι διαπραγματευτικέ ομάδε. Δεν πρόκειται για ένα εναλλακτικό κείμενο. Απλά ουσιαστικά θέλουμε να σας δώσουμε και εμείς τις δικές μας εμπειρίες για να σας πω πώς θα γίνει, θα συγκρίνουμε ε, άρθρο προς άρθρο τα διάφορα κείμενα Συμβουλίου Επιτροπής, ε, το προτινόμενο έγγραφο για να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες και μετά τη μεταρρύθμιση. Δεν θέλουμε να ε, γίνουν πιο αδύναμες ε, οι ε, εγγύησεις και οι διασφαλίσεις. Θέλουμε να υπάρχει επίσης τα επόμενα χρόνια ένα ευέλικτο προσανατολισμένο προς το μέλλον σύστημα, κατάλληλο της μικροπιστής επιχειρήσης, ουδέτερο τεχνολογικά. Δεν θέλουμε να υπάρξει γραφειοκρατία, ιδίω για τους νέους δεκανισμούς και ρυθμίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων φορέων εποπτείας. Θα πρέπει να ε, ε, λειτουργήσει και το one-stop shop, αλλά και οι λεγόμενοι μηχανισμοί εγκύτητας. Απλή νόμη, γιατί αυτή είναι και πιο αποτελεσματική. Αυτό που επίσης μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τις νέες τεχνολογίες. Η μαζική συλλογή δεδομένων είναι ένα γεγονός και είναι αποτέλεσμα απογραφής ε, πολλών δεδομένων, ε, εντοπισμός κάποιων ε, ιστοσελίδων μηχανών αναζήτησης. Εμείς θέλουμε και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, στην ιδιωτική σφαίρα, να γίνει σεβαστό, γιατί είναι και στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης είναι μια σημαντική αρχή. Προσπαθούμε λοιπόν αυτές τις νέες τεχνολογίες να τις αξιοποιήσουμε τρόπο που να μην ε, θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των ε, ατόμων. Θέλουμε να δούμε και τι ηθικές δεντολικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν οι νέες τεχνολογίες. Τι σημαίνουν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες για τα επόμενα χρόνια. Καλώς ε, λοιπόν λόγος αυτός για να ολοκληρώσουμε αυτό το έγγραφο με ένα position paper που όπως σας είπα ε, θα συμπληρώνει κάποια στοιχεία. Και ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας θέλω να αποτέσω φόρο τιμής στον Πίτερ Χάστινγκ, στον προκάτοχό μου. Μας ενέπνευσε για πάνω από 11 χρόνια ως επόπτης, ως σύμβουλος ε, ε, πήρε τον οργανισμό μας από τα σπάργανα και τον ορίμασε. Θέλουμε τώρα να δείξουμε ηγεσία για να κάνουμε θετική διαφορά στις ζωές των απλών πολιτών. Βασιζόμενοι στην εμπειρία και του Πίτερ. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας. Και αγαπητέ Πρόεδρε, να σας δώσω συμβολικά και ένα αντίγραφο της ε, ετήσιας έκθεσης. Παρακαλώ, εκ προσωπικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, κ. Μπουτελή, γιατί θα πρέπει να φύγει σε 30 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ζητήσω να τηρήσετε τα χρονικά όρια, να είμαστε σύντομοι στα σχόλιά μας. Ο κύριος είναι πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αιτήσια αυτή έκθεση. Νομίζω ότι είναι καλή η χρονική στιγμή για να εκφράσουμε ποιες είναι οι νέες προκλήσεις οι οποίες είναι κοινέ και για την Επιτροπή Λίμπε, για το Κοινοβούλιο, αλλά και για τη δική σας υπηρεσία. Καταρχάς, πώς ε, μπορείτε να μας υποστηρίξετε κατά τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου. Ξεκινήσαμε τον τριγωνικό αυτό διάλογο για το TPDR και νομίζω ότι η γνώση σας από πλευράς της υπηρεσίας σας είναι πάρα πολύ σημαντικές για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να πλουστεύσουμε κάποιες λύσεις σε ε, ναι ή όχι και πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη δική σας την παρέμβαση και την συμβολή ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική για το σχέδιο εφαρμογής, κλειδί για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Και αυτό επειδή πιστεύω ότι δεν τελειώνει η δουλειά φέτος. Θα πρέπει να κάνουμε σκληρή δουλειά με όλες ε, τις εθνικές υπηρεσίες της χώρας του καθενός. Αυτό λοιπόν θα σας απασχολήσει και εσάς. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε εσείς και η υπηρεσία σας στο σχέδιο εφαρμογής και στην προώθηση της ε, γνώσης, την ευαισθητοποίηση για το θέμα της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τα καινούργια φαινόμενα, γιατί ξεκινάμε τη συζήτηση για την ψηφιακή κοινή αγορά στην Ευρώπη και νομίζω ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν ε, εντελώς ε, νέες ε, προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη ρομποτική, το εμπόριο, την υγεία. Ποια είναι λοιπόν η συμμετοχή σας και η συμβολή σας για το δικό μας το έργο στο μέλλον. Και τελευταίο σημείο, γιατί δεν θέλω να ακρηγορήσω. Πείτε μας τι πιστεύετε. Και ποια είναι η άποψή σας για την οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα, το e-privacy. Αυτό θα πρέπει να είναι επιπρόσθετο προς το έργο της προστασίας των δεδομένων. Ευχαριστώ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπουταρέλη, δεν θα σχολιάσω την ίδια την έκθεση. Δεν είχα χρόνο να τη διαβάσω προσεκτικά. Αλλά, όπως ξέρετε, είναι πολύ καλή εντύπωση ε, της υπηρεσίας σας, του έργου της υπηρεσίας σας. Και το ίδιο ίσχυε και για τον κύριο Hastings που ήταν πολύ καλός επόπτης και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα είσαστε πολύ καλό καλός επόπτης ε, προστασίας δεδομένων. Θα αναθεωρήσουμε το έργο σας του χρόνου. Ο, ο συνάδελφος έθεσε διάφορα ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για την δουλειά που έχει γίνει από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον κανονισμό, στα πλαίσια του κανονισμού και τη οδηγία. Σχολιάστε παρακαλώ τρει τομεί. Καταρχάς, ποια είναι η άποψή σα για το αποτέλεσμα τη νέα νομοθεσία. Κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση. Ή μήπως ε, διακινδυνεύουμε να μειωθεί το επίπεδο της ε, προστασίας. Είπατε ότι θα θέλατε μεγαλύτερο επίπεδο, υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Πιστεύετε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Δεύτερη ερώτηση. Για τη διαδικασία. Όπως ξέρετε, το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο εξ αρχής ήθελε να αντιμετωπιστεί το, η συμφωνία αυτή ως πακέτο, η οδηγία και ο κανονισμός το Συμβούλιο δεν μας προκάλεσε έκπληξη, προτιμούσε να δεχτεί τη συμφωνία για τον κανονισμό πιο πολύ από ότι για την ε, οδηγία. Και πολύ φοβάμαι ότι θα ξανανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου. Για να μην προκαλέσουμε ρήξη στις διαπραγματεύσεις. Να συμφωνηθεί δηλαδή πρώτα ο κανονισμός και μετά η οδηγία. Τι πιστεύετε γι' αυτό. Τρίτον, σχολιάσατε το νέο εργαλείο. Δεν το κατάλαβα ακριβώς αυτό που είπατε. Τι λέτε ότι το εργαλείο αυτό θα μας βοηθήσει στους δρεμερείς διαλόγους ή ε, μήπω μιλούσατε για κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Καταρχά, θα ήθελα να υποδείξω το εξή. Επειδή υπάρχουν ε, ακριβώς αυτές οι εξελίξεις ε, στην ψηφιοποίηση, χρειαζόμαστε πιο υψηλά επίπεδα προστασίας για την προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής σφαίρας και θα ήθελα να Αναφέρω μια πρόταση από έναν ανακοινωθέν τύπου σας όπου λέτε ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων που ισχύει σήμερα λέει ότι η γνώση εξυπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο, αλλά κάποιες φορές μου δίνεται η εντύπωση ότι η τρέχουσα συζήτηση όπου μιλάμε για την ψηφιακή αγορά κινούνται αντίστροφα. Γιατί Μιλάμε για τις ευκαιρίες για την αγορά, για τις επιχειρήσεις, όχι όμως για το ερώτημα του τι θετικό αντίκτυπο θα έχει αυτό για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, γιατί οι πολιτικοί και πολλοί πολίτες στην παρούσα φάση πιστεύουν ότι δεν πειράζει ε, να γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα για μένα, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Όσο πιο πολλά όμως στοιχεία συλλέγονται, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμο ότι δεν έχει σημασία τόσο πολύ το κάθε στοιχείο, το κάθε δεδομένο από μόνο του, αλλά το profiling που γίνεται. Η ανάλυση οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων έχει συνέπειες. Μπορεί να έχει καλές συνέπειες και να χρησιμοποιείται για καλούς σκοπούς, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και αρνητικός αντίκτυπος, για παράδειγμα για πιο ακριβές ε, ασφάλειες, ε, για να μην πάρει κάποιος ε, δάνειο, ανυπόθηκο, γιατί θεωρείται κακός πελάτης και ενδεχομένως να αποκλείεται και από κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η προστασία των δεδομένων. Και σήμερα διάβασα στις ειδήσει ότι το PayPal ενδεχομένω να μην είναι τόσο καλό όσο φαίνεται, γιατί ω τώρα όλοι θεωρούν ότι είναι γρήγορο και καλός και ασφαλής τρόπο πληρωμής μέσω του διαδικτύου του PayPal. Αλλά σήμερα διάβασα ότι άλλαξαν οι όροι στο PayPal και όταν χρησιμοποιεί κανείς ουσιαστικά δίνει το όνομά του τη φωτογραφία τα στοιχεία του λογαριασμού του, οτιδήποτε έχει εκεί. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για όποιο σκοπό θέλει. Και το μοναδικό που μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι να μην τα χρησιμοποιήσει πολύ απλά. Και αυτό ίσως για κάποιους είναι καλύτερο, γιατί ε, ίσως να είναι προτιμητέο να αγοράζει κανείς για παράδειγμα ένα βιβλίο στην τοπικό βιβλιοπωλείο και όχι ε, στο διαδίκτυο. Αλλά αυτό λοιπόν αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση του πακέτου προστασία δεδομένων, αλλά χρειάζεται ένα πακέτο το οποίο θα πληρεί όλα τα κριτήρια. Ευχαριστούμε, Μπίρκιτ. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην επαναλάβω αυτά που ακούσαμε ήδη για που είπε ο κύριος Σοϊκοέλιο, η κυρία Σίπελ και άλλοι συνάδελφοι, γιατί εγώ θέλω να ακούσω πραγματικά τις απαντήσεις σας στα σημεία αυτά, τα οποία μας απασχολούν και εμάς. τέρος, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας για τις συζητήσεις που γίνονται για το κείμενο του κανονισμού. Είναι περίεργος λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για τις ισχυρισμούς ότι οι θέσεις αυτές του Κοινοβουλίου και, της, ε, και του Συμβουλίου μπορεί να παρεμποδίσουν και την ανάπτυξη. Θα ήθελα να ακούσω την απόψή σας. Αν συμφωνείτε, ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση μεταξύ της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της δυνατότητας επεξεργασίας δεδομένων για πιο πολλές ε, πληροφορίες. Ή μήπως θεωρείτε ότι υπάρχει μία αλληλεξάρτηση. Και δεν αυτό αποκλείονται. Γιατί αυτό προφανώς είχαν κατά νου τα κρατημέλη και οι πιο πολλοί βουλευτές εδώ όταν κατάρτισαν το κείμενο της ε, μεταρρύθμισης. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε μια τέτοια συζήτηση γιατί έχω την αίσθηση ότι απομακρυνθήκαμε κάπως από αυτή την αρχή. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι ή το ένα ή το άλλο. Και όχι ότι τα δύο αυτά θα πρέπει να κινηθούν εκ παραλλήλου. Και πώς μπορούν από τεχνικής άποψης να συνάντουν αυτές οι δύο αρχές. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα επίσης να μου πείτε το πώς αξιολογείτε την τρέχουσα συζήτηση για την αναλογικότητα της χρήσης προσωπικών δεδομένων για την ασφάλεια γιατί όπως ξέρετε στα κρατημέλη ακόμα συζητάμε το θέμα τα φύλαξη προσωπικών δεδομένων και τηλεπικοινωνιών και συζητάμε επίσης ε, τα, την φύλαξη των ε, δεδομένων επιβατών και ξέρω ότι η έχει ο Ευρωπαίος ε, έχει καταρτήσει σχετική έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας για το θέμα αυτό και το πώς μπορούμε να πετύχουμε πιο πολύ εναλλαγικότητα σύμφωνα με αυτά που είπε και το δικαστήριο πέρσι. Έχετε κάποια συμβουλή να μας δώσετε από τις δικές σας αναλύσεις από την τελευταίο χρόνο μετά τη λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ κυρία Άννα Γκόμες. Σας ευχαριστώ κυρία Μπουταρέλη. Να ρωτήσω αν παρακολουθήσατε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, τις διαπομοτεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την προστασία δεδομένων και συγκεκριμένα υπό το φως των αλλαγών που οι Αμερικανοί σκέφτονται να κάνουν ώστε να υπάρχουν ένδεικα μέσα και δικαστική, δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για τους Ευρωπαίους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στον ιδιωτικό βίο και της προστασίας του. Σας ρώτησαν για τη συμφωνία αυτή ελεύθερου εμπορίου και απελευθέρωση των υπηρεσιών στα πλαίσια του ΠΟΕ. Διότι από ό,τι ακούω για τις συμφωνίες αυτές ουσιαστικά απορριθμίζει τον τομέα των υπηρεσιών καθώς είναι ένας τομέας όπου ο έλεγχος των δεδομένων είναι ζωτική σημασίας. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε που έχετε φτάσει και η ερώτησή μου, ο ρόλος σας, είναι να ασχολείστε και με την επιβολή του νόμου και την επικοινωνία και την ενημέρωση και την λεπίδραση με τις εθνικές αρχές. Πώς εξελίσσεται αυτή η συνεργασία. Εγώ ανησυχώ για τη χώρα μου όπου ο η εθνική μας αρχή ετοιμάζει υπέροχες εκθέσεις όπου τονίζει πολλά από τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν στην νομοθεσία ή στην πράξη και η Εθνική μας Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων γιατί μια πολύ ωραία έκθεση που ανέφερε ότι η εφαρμογή του ΦΠΑ γινόταν με τρόπο τελείω που συμπίπτει με, μορφή διακριτικής μεταχείρισης Φαίνεται τελικά ότι οι εταιρείε, οι συμβουλοί του ε, και οι υπηρεσίε του μπορεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ε, φορολογουμένων μέσα από τι εφορίε. Δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι ιδιαίτερα παραπλανητικό ή βλαβερό για του φορολογούμενου. Έχει γίνει κάτι γι' αυτό, διότι η αρχή προστασία των δεδομένων μα σε εθνικό επίπεδο δεν είχε τοποθετηθεί ω προ αυτό το θέμα. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν ω προ την επιβολή. Ευχαριστούμε. Μαριού. Ευχαριστώ κύριε Μπουταρέλη για την ε, έκθεση. Το πιο ενδιαφέρον τμήμα ήταν οι ε, στόχοι για το 2015 και εξής. Οι σκιώδεις και ομάδες τους ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το εργαλείο που θα μας δώσετε, γιατί ήδη έχουμε τριμερή διάλογο και από το 2014 έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε το κείμενο. Έχετε αργήσει λοιπόν κάπως και πραγματικά ευνηδιάστηκα, διότι δεν ανήκουμε στην γενιά Z που ε, αναφέρατε και θα χρησιμοποιούσε μια εφαρμογή στο κινητό. Δεν θα μας βοηθούσε πολύ σε αυτές τις συνθήκες, οπότε ίσως να είχαμε μια μορφή πιο αποτελεσματική για να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Ως προς τη ρύθμιση και όλα αυτά τα στοιχεία που αναπτύσσεται, που συγκεντρώνεται μάλλον για τις μεγάλες προκλήσεις, τον ε, υπολογιστική νέφου, το, ε, τα μεγάλα δεδομένα, πιστεύετε ότι λείπει κάτι από την αλυσίδα πληροφορησής μας λόγω χάρη την κοινή ευθύνη του παρόχου και του ε, διάμεσου εφόσον είναι ένας χώρος λόγου χάρη στην ε, αν είναι ένας χώρος στο υπολογιστικό νέφος, πρέπει να τους αφήσουμε να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. Ε, θα ανοίξουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία για το μέλλον. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω εσείς προηγείστε λίγο στις, ε, στην εξέταση του θέματο από εμά. Αλλά τι σκέφτεστε, υπάρχει μεγάλο κενό που πρέπει να καλυφθεί, μικρότερο, πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να το υπερβούμε. Και η τρίτη ερώτησή μου για τις ε, επικοινωνίες διασύνδεσης και την εκπαίδευση. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο, διότι υπάρχει πολλή εκπαίδευση για τους ειδικού, ε, τους εξειδικευμένους ανθρώπους. Αλλά αν μιλήσουμε για τους καταναλωτές και τις νεότερες γενιές ή και τις μεγαλύτερες. Δεν έπρεπε να επεξεργαστούμε μια γενική προσέγγιση για να βλέπουμε τα βιογραφικά στα σχολεία διότι τα εθνικά κράτη θα μου πείτε το ρυθμίζουν αυτό, όμως έχουν πολύ διαφορετικές θέσεις για, την, για τον ψηφιακό χώρο τα εθνικά κράτη. Δεν θα ήταν καλό όλες οι χώρες να, έχουν, να δίνουν ίδιες ευκαιρίες, την ίδια δυνατότητα να αναπτύξει κανείς μια ψηφιακή υγιεινή. Ποιος είναι ο ρόλος σας αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα κύριε Μπουταρέλη έχετε το λόγο για να κάνετε τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας για αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα έπρεπε να μείνω κάμια δυο μέρες για να τα πούμε όλα. Οπότε θεωρώ ότι με καλείτε ξανά στην ουσία. Κύριε Μπόρνη, για να ξεκινήσω με την ερώτησή σας. Θα θέλαμε σήμερα να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο. Όχι όταν θα είναι πολύ αργά. Είμαστε ανεξάρτητοι αρχή δεν διαπραγματευόμαστε, δεν είμαστε επισήμω μέρος κανενό τριμερού διαλόγου. Είμαστε όμως ο άμεσος βασικός σύμβουλος των ε, σχεδιαστών της νομοθεσίας και της Επιτροπής. Θέλουμε σήμερα να δράσουμε ε, ως ε, υπεύθυνοι για τις λύσεις που θα βρεθούν και τα προβλήματα. Και να προλάβω και μια από τις επόμενες ερωτήσεις απαντώντας αυτό. Αν με ρωτήσετε στην 23η χρονιά όπου εργάζομαι για την προστασία δεδομένων σε διαφορετική θέση ίσως. Δεν είναι αυτή η ιδανική μεταρρύθμιση για μένα. Έχω ετοιμάσει πολλές εθνικές διατάξεις και έχω προτείνει πολλές τέτοιες και ίσως αν το ξαναέκανα δεν θα ακολουθούσα ακριβώς τις σημερινές προτάσεις. Όμως τα πράγματα στη ζωή είναι περίπλοκα και πρέπει να παραμένουμε στο κείμενο που τώρα ε, μας προσφέρεται. Δηλαδή, το βασικό είναι να εμποδίσουμε τον νομοθέτη να διαπράξει σφάλματα. Διότι το επαναλαμβάνω το μήνυμα αυτό μα και τέλο ο κόσμο, όλοι περιμένουν μια τέλεια διέξοδο. Αλλά δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε διέξοδο είναι και κακή. Γι' αυτό περιμένουμε την απόφαση για την οδηγία από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση το κείμενο που θα συνταχθεί τον Ιούλιο θα συμπληρωθεί από εμάς ως το Σεπτέμβριο ως προς τις ιδεολογικές σκέψεις ε, εκτιμώντας θα τοποθετούνται θετικά και όχι αρνητικά και θέλουμε όλη αυτή η διαδικασία να γίνει γέρος για την οδηγία. Πρέπει να περιμένουμε όμως για το κείμενο του Συμβουλίου πρωτού ε, ξεκινήσουμε να δίνουμε τις προτάσεις μας. Το τελικό κείμενο θα το έχουμε τον Ιούνιο για το εκτελεστικό σχέδιο. Πολύ δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα. Περιμένουμε η μεταρρύθμιση να εγκριθεί για τρίτη φορά από το Συμβουλίο, όπως επαναλήφθηκε συχνά στη συζήτηση 25 και 26 Ιουλίου φέτος, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να εγκριθεί επισήμω 28 γλωσσικές εκδοχές, για να γίνει σύγκριση μεταξύ του, για να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα, για να τεθεί σε ισχύ. Τον Ιούνιο-Ιούλιο του χρόνου. Οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και υπάρχει περιθώριο ελιγμών για τη μετάβαση, αλλά για ποια μεταβατική φάση ε, μιλάτε, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Προστασία των Δεδομένων θα ξεκινήσει και τι θα γίνει με τις κατεξοδότηση και τις κριτικέ πράξει. Νομίζω την απάντηση πρέπει να τη δώσουμε με ήπια νομοθεσία. Δηλαδή συστάσεις, κατευθυντήρες γραμμές, πρακτικέ πρακτικές, ε, αρκετά ευέλικτε, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στι ανάγκε μα, Αλλά με πιο ε, επιλεκτική και ισχυρή και αποτελεσματική αρχή προστασία των δεδομένων. Η Επίτροπο Γιούροβα, την οποία συνάντησα μόλι πριν από εσά, θέλει να συνεργαστεί μαζί μα. Για να επιτρέψει στην αρχή μα, επειδή δίνουμε συμβουλευτική και στι υπηρεσίε στην γραμματεία τη να αναλάβει πλήρω το καθήκοντά τη. Πρέπει να επιτρέψουμε στου συναδέλφου να ορίσουν την αρχιτεκτονική που θέλουν, να εργαστούν επιλεκτικά, διμερό να ασχοληθούμε με πολύ επιλεγμένες υποθέσεις, διότι ασχολούμαστε με 12-15 υποθέσεις το χρόνο. Και αν ασχολούμαστε με τέτοιες υποθέσεις τώρα, είναι όχι απλώς επειδή έχουμε μεγάλο φόρτο εργασία, αλλά επειδή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο. Κάτι που θα το διατηρήσουμε και στο μέλλον. Πέραν του συμβουλευτικού ρόλου, η αρχή πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Η ερώτησή σας για τα νέα φαινόμενα. Οι νέε αυτές προκλήσεις, όπως είπα για τη στρατηγική μας, είναι προκλήσεις που θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε ως μια ανεξάρτητη αρχή με ε, νέες τεχνολογίες γιατί η αριστεία μας δεν αφορά μόνο την προστασία των δεδομένων, αλλά και την επιβολή του νόμου με ψηφιακά μέσα. Σύντομα, η ομάδα κρούσης θα ασχοληθεί με την IT, ITP και οι δουλειές μας στο δίκτυο ήταν τόσο τα αποτελέσματα μας στο δίκτυο ήταν τόσο θετικά που θα οργανωθεί και η επόμενη φάση σύντομα με αυτή την οπτική γωνία πρόθεσή μου είναι να έχουμε στο, στην ε, Silicon Valley μια μακρά επίσκεψη όχι για να, συζη... να συναντήσουμε μόνο τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών, αλλά για να μιλήσουμε με τους ερευνητέ, τους ε, ε υπεύθυνου, όσους λαμβάνουν τις ιδέες, να μας εμπνεύσουν, να δούμε πώς θα είναι πιο αποτελεσματικοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες με όλα τα δεδομένα υπόψη. Και ω προ την ερώτησή σα για τον ιδιωτικό βίο, είναι απλό. Πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι αργά να γίνει με τη μεταρρύθμιση αυτή. Αλλά υπήρξε δέσμευση να γίνει σε δύο φάσει αυτό και εκτιμώ την πρόθεση αυτή. Είμαι πρόεδρο τη ομάδα εργασία που το 1996 ε, συνέταξε το πρώτο σχέδιο πρόταση για την ε, οδηγία για τι τηλεπικοινωνίε. Τώρα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει πλήρη συνέπεια μεταξύ των δύο ξέρω ότι μια ομάδα ζητά τελευταία στιγμή αλλαγέ στην οδηγία, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά ποιε είναι οι ανάγκε μα και νομίζω ότι η οδηγία πρέπει να αντικατασταθεί από διατάξει κανονισμού. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να δίνουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη και περιθώριο τα στα μελη Κύριε Κοέλιου, νομίζω το νομικό πλαίσιο που θα προβλέψουμε θα πρέπει να είναι πιο ισχυρό και πιο εύρωστο για να μπορεί να αντισταθεί σε αυτές τις τεχνολογίες. Η άποψή μου για τη δουλειά που έχει γίνει σήμερα ε, είναι αν είμαστε στον ορθή ή όχι πορεία. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Υπάρχει ακόμη περιθώριο. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο κάποιες διατάξεις, ιδίως η αρχή περιορισμού και των νόμιμων συμφέρων, πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση. Υπάρχει κίνδυνος να ελαχιστοποιήσουμε κάποιες διασφαλίσεις ή να ε, παραμένει πολύ περιθώριο σε εθνικό επίπεδο. Για την πρόληψη των κλίματος ξέρουμε ότι πρέπει να, ε, ασχολη... να καλύψουμε το θέμα αυτό ξεχωριστά στην οδηγία από ότι για την επιβολή. Η πρόθεσή μου είναι η συζήτηση αυτή να είναι διαφανής. Όχι για το δικό σας μονόφελος, αλλά για τον καθένα στον κόσμο Πρέπει να καταλαβαίνει σήμερα τι κάνουμε για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Και βεβαίω πρέπει να υπάρξει κάποιο πακέτο. Σωστά το Συμβούλιο αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτά ως δέσμη μέτρων και ως τέτοια πρέπει να την ε, μεταρρυθμίσει με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων. Με ρωτήσατε κυρία Γκόμες που είμαι και σας είπα στη σωστή πορεία. Αλλά πρέπει να εξυγχρονιστούμε σύντομα και να επιτρέψουμε σε αυτά τα εργαλεία να τεθούν σε ισχύ την ίδια στιγμή. Όχι όπως έγινε το 2004 για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς. Έχουμε ε, Παφέ για τι μεγάλε κλίμακες βάσει δεδομένων και τι περιοχέ του τρίτου πυλώνα όπου παρακολουθούμε κάποιε από τι δράσεις τη Επιτροπή. Μιλώ για τις βάσεις δεδομένων που έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και από τα κάτι μέλη το ίδιο. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με βάση κοινού κανόνε. Αυτά δεν θα γίνουν όλα σήμερα. Η εφαρμογή θα είναι μια ευκαιρία να υπάρχει ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να μεταφέρει κανεί παντού. Κυρία Λόριστη, να είστε βέβαιοι ότι θα σα δώσουμε όλε τι επιγραμμικέ διευκρινήσει που χρειάζονται και για τον ιστότοπο, αν χρειαστεί και επιθάρτου. Αλλά δοκιμάσαμε την ε, εκδοχή αυτή και θα επιτρέψει λόγω χάρη σε δύο δευτερόλεπτα να μπορεί κανεί να δει που υπάρχουν ε, παγίδε στο κείμενο τα δεδομένα υγείας, γενετικής, οτιδήποτε. Κυρία Σίπελ, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Να σας αναφέρω το αποτέλεσμα του Ευρωβαρομέτρου, της μελέτης του Ευρωβαρομέτρου το, από τον Ιούνιο φέτος, 20 χρόνια μετά την, εισαγωγή της, την θέση και της οδηγίας το 1995, Μόνο μια μειονότητα δηλαδή, 15% αισθάνονται ότι ελέγχουν πλήρως τα δεδομένα τους. 20 χρόνια μετά την ε, θέση σε ισχύ της βασικής οδηγίας. Ως προς την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, καθημερινά αναγκαζόμαστε να παρέχουμε τις πληροφορίες μας. 71% των ανθρώπων θεωρούν ότι πρέπει να το αποδεχτούν. Να αποδεχτούν την εναλλακτική που προσφέρεται. Και ένα στους 10 ένα στους δέκα λέει ότι ενημερώνεται παρκώς για τη συλλογή πληροφοριών. Θα μιλήσουμε ειλικρινά λοιπόν. Μπορεί να δυσαρεστήσουμε κάποιους από τους νομοθέτες, αλλά επειδή και λογοδοτούμε και είμαστε ένα οργανισμό επαγγελματιών, θέλουμε να επικεντρωθούμε στην αλήθεια. Κυρία τα μεγάλα δεδομένα χρειάζονται και μεγάλη προστασία. Πολλές φορές στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε τις ίδιες δυσκολίες. Η προστασία δεδομένων δυσκολεύει την κοινοτομία και ανάπτυξη. Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε τα ευεργετικά αποτελέσματα των μεγάλων δεδομένων, αλλά η καινοτομία και η ανάπτυξη μπορούν να υπάρξουν μόνο εφόσον, έχουν ένα, μόνο εφόσον υπάρχει εύρωστο σύστημα προστασίας του βίου. Για σκοπούς αναλογικότητας θα σας υποκληθεί μια πρόταση για το 43α για την παρακολούθηση θεωρούμε ότι η οδηγία της ηλεκτρονικής του ηλεκτρονικού ιδιωτικού βίου και το άρθρο 15 είναι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για κάθε εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια. Κυρία Γκόμες, για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών χθες είχαμε ένα σημαντικό εργαστήριο για τα δικαστικά για, τα δικαστικά, για τις δικαστικές προσφυγές. Έχουμε καλά νέα για τις ΗΠΑ αλλά υπάρχουν και όρια. Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν υπάρχει μόνο μία ιδέα. Χρειάζονται βελτιώσεις για το TTIP. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε, κατά την άποψή μας. Η προστασία των δεδομένων πρέπει να παραμένει στο κέντρο της μεριμνάς μας και ο ρόλος ε, παρακολούθησης και ελέγχου που ασκούμε βελτιώνεται πολύ. Είμαστε ικανοποιημένοι με το τωρινό επίπεδο για την ε, γνώση περί προστασίας των δεδομένων που υπάρχει, αλλά η λογοδοσία πρέπει να γίνει ακόμη πιο έντονη και η προστασία των δεδομένων ακόμη πιο εύρωστη και αυτή και αποτελεσματική. Ε, κυρία Λόρεστιν, και εδώ θα κλείσω νομίζω. για την ανάληψη ευθύνη και για τον έλεγχο των παρόχων. Θα τα δείτε στην έκθεσή μα. Τα μελετήσαμε πέρσι για την υπολογιστική νέφου και για το ποιο είναι υπεύθυνο για ποιο πράγμα. Και τη συνένεση. Διότι οι άνθρωποι, οι πολίτε τώρα δεν. Ε, μάλλον οι άνθρωποι αυτοί δεν νοιάζονται για το ποιο είμαστε. Ποιοι είμαστε. Θέλουν τι προτιμήσει μα να ξέρουν. Πού βρισκόμαστε, τι μα αρέσει αλλά ουσιαστικά κάνουν, ε, βγάζουν κέρδος από αυτό γνωρίζοντας τις ε, βασικές ανάγκες του ιδιωτικού μας βίου. Θα συμφωνήσω με την κυρία Γιούροβα που μόλις είδα πριν από ένα μισάωρο. Θα συνεργαστούμε σε όλη αυτή την προσπάθεια ώστε να ε, εισαχθούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μόλις γίνει η μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί, μαζί μας. Our next item Επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι το σχέδιο γαλλικού νόμου για την παρακολούθηση. Έχουμε ένα θέμα με τη συμβατότητα αυτού του νομοσχεδίου με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα θέλαμε να δούμε και τα περί προστασίας δικαίου, μηχανισμό φύλαξης δομένων, δικαιώματα των ε, προσώπων κτλ. Επειδή είναι θέμα το φύλακα ε, των συνθηκών οικομισιών, χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μα τον κύριο Φρανθίσκο Φωνσέκα Μωρίο, Διευθυντή Ποινική Δικαιοσύνη τη Επιτροπή, που θα μα παρουσιάσει την άποψη τη Κομισιόν για τον νέο αυτό γαλλικό νομοσχέδιου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή... In this, uh, uh, committee, the opinion of... Σας ευχαριστώ λοιπόν με τον ε, Επίτροπο Τίμερμαν και την Επίτροπο ε, Γιουροβά ασχολούμαστε με το θέμα της μαζικής παρακολουθήσης γενικότερα, αλλά θέλετε να συζητήσουμε σήμερα τον γαλλικό νόμο για την παρακολούθηση. Επειδή είναι ε, γαλλικό θέμα αυτό, ας μιλήσω γαλλικά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι σημειώνουμε τα δύο, τις δύο επιστολές που στείλατε ορισμένοι εξημών προς τον κύριο Τίμερμαν, στην Επίτροπο Γιώργα, στον Επίτροπο Αβραμόπουλο και την γραπτή ερώτηση σημειώνουμε, την οποία καταθέσατε. Απάντησε πριν από μια εβδομάδα ο Αντιπρόεδρος Τίμερμας στην επιστολή αυτή. Σημειώνουμε λοιπόν τις ανησυχίες της Επιτροπής σας σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Καταρχάς αυτό. Κατά δεύτερον, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα, διότι η παρουσία μου εδώ ανεξαρτήτως των τεχνικών, νομικών, διαδικαστικών ζητημάτων, σεβασμού, εγγύσεων κτλ. Δείχνω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την κατάσταση αυτή Πιθανή παρέμβαση, ε, παρεμβατισμού στην ιδιωτική ζωή, πιθανής επαναλαμβάνω, δεν έχει ακόμη εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο, σε περιπτώσεις όπως αυτή που μας απασχολεί σήμερα. Όμως, αν μου επιτρέπετε, θέλω καταρχά να σας πω ότι όλοι γνωρίζουμε και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν ποια είναι η πολιτική, θεσμική, δημοσιονομική, συγγνώμη, διαδικαστική κατάσταση σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό το οποίο εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου από την Άνω και κάτω Γαλλική Βουλή. Πρέπει όμως να είναι σαφές το εξής. Και αν δεν απατώμε στα ζητήματα του Γαλλικού Συνταγματικού Δικαίου, εγκρίθηκε, αλλά δεν έχει τεθεί σε ισχύ αυτό ο νόμος ακόμη. Δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει εγκριθεί, γιατί υπήρξε προσφυγή από 100 τουλάχιστον ε, Γάλλους βουλευτές ε, στο συνταγματικό ε, συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα από πολιτική πλευρά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, και θα με διορθώσετε αν κάνω λάθο, για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γαλλική Δημοκρατία, ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία αποφασίζει να συνταχθεί με του βουλευτέ που κατέθεσαν την προσφυγή στο Συνταγματικό Συμβούλιο. Και τώρα έρχομαι στο πρώτο μου συμπέρασμα, αν θέλετε, σε πρώτη μου διαπίστωση θεσμικού χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα πιστεύω, 2 Ιουλίου, πρέπει να αφήσουμε πρώτα απ' όλα να μιλήσει το Συνταγματικό Συμβούλιο. Σε, γιατί πρέπει να σεβαστούμε το κράτος δικαίου στη χώρα. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ικανοποιητική απάντηση αυτή. Είμαστε ακόμη όμως σε μια πολύ σημαντική φάση, διότι ο βασικός θεματοφύλακας της ενταγματικότητας του νόμου δεν έχει αποφανθεί ακόμη. Σίγουρα είχαμε την ευκαιρία να φιλομετρήσουμε και να δούμε αυτό το νομοσχέδιο, γνωρίζουμε βεβαίως τι είπε και ο επόπτης δεδομένων για την αναλογικότητα κυρίως, αλλά εμείς πρέπει να σεβαστούμε αυτό που θα πει ο βασικός θεματοφύλακας στη Γαλλία, δηλαδή το συνταγματικό Συμβούλιο. Όμως, και περνάω στα αγγλικά τώρα, να τονίσω το εξή. Όλοι γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση. Της 23 Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος Τιμερμάν σας απήντησε επισήμως σε γραπτή ερώτηση για τα δεδομένα. Και η δική μου αρχή δήλωσε τα εξής. Η ερώτηση των ε, αξιότιμων ευρωβουλευτών εγείρει σημαντικά νομικά θέματα. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι το γεγονός αυτό. Κατά δεύτερον, και συνεχίζω να διαβάζω, βάσει των ε, ε, συνηθισμένων πρακτικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει για την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους εφόσον υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί βάσει του νόμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η επίσημη γραμμή μου. Και πρέπει να την επαναλάβω εδώ. Το μόνο για το οποίο μπορώ να σας καθησυχάσω και που μπορώ να σας πω είναι είναι ότι θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Βάσει μιας θεμελιώδους αρχής. Ισορροπία μεταξύ θεμελιώδων δικαιωμάτων και ασφάλειας. Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Ευρώπη αναγκάζει τα κράτη-μέλη ως περίσταση να βεβαιωθούν για την ασφάλεια των πολιτών. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ χωρίς να υπάρχει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η βασική μας πολιτική γραμμή, όπως έχει καταρτιστεί στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια. Την, στην πιο πρόσφατη εκδοχή, εκδοχή που γνωρίζετε πολύ καλά. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει με το θέμα αυτό, όπως θα έλεγα οι Γάλλοι με μια έκφρασή τους. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα τους ε, θεματοφύλακες των ε, νόμων και την άποψή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας αυτή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο μέλη της Επιτροπής. Η ε, κυρία Γκρίσπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μωρίγιο για την παρουσίαση αυτή στην οποία βρίσκουμε την περιβόητη το περιβόητο διπλωματικό και νομικό του ταλέντο και ικανότητα. Είναι ένα νομικό κείμενο αυτό που δημιούργησε κάποιες απορίες σε κάποιους ευρωβουλευτές. Στη φάση της συζήτησης Ακόμη δηλαδή και όταν ήταν νομοσχέδιο. Εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου βέβαια. Δεν έχει αναχθεί σε νόμο ακόμη. Αυτό προβλέπεται και εξαρτάται από την απόφαση την οποία θα λάβει αφού το επιλήφθηκε το Συνταγματικό Συμβούλιο. Μετά από προσφυγή βουλευτών, όπως βλέπετε, και με τον πρόεδρο της αυτή τη φορά. απάντησε η Επιτροπή επισήμως ερωτήσεις μας. Να σας ε, πω κάποια πράγματα πιο δεξοδικά μετά πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά το ζήτημα είναι, ε, έχει να κάνει με το σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας ε, και αν συνάδουν οι διατάξεις αυτές με το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείτε να απαντήσετε απόψε όμως μας είπατε γιατί υπάρχει αυτή η προσφυγή του Συνταγματικού Συμβουλίου που ουσιαστικά αναστέλει και την ε, έκδοση του νόμου και τη δική σας απάντηση. Θέσαμε πάντως ε, εμείς ε, ερώτημα στην Κομισιόν, πήραμε απάντηση από τον Αντιπρόεδρο Τίμερ μας, αναφερθήκατε. Δεν ξέρω όμως αν τα κατάλαβα όλα καλά όπως τα είπατε, αλλά η απάντηση ουσιαστικά θέτει, πώς να το πω, αναφέρει τέλος πάντων το ενδεχόμενο να ε, εγείρονται σημαντικά νομικά ζητήματα. Ε, είναι λίγο συμβιλικό κάπως αυτό, ως απάντηση, αλλά μας δημιουργεί ε, τις απορίες αυτές για το κατά πόσο είναι συμβατό αυτό το νομοσχέδιο. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι μου φαίνεται και κατεπήγον και απαραίτητο και επιτακτική ανάγκη να δοθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο στη Γαλλία σε ό,τι αφορά την συλλογική χρήση δεδομένου. Τέλο πάντων να βγούμε από αυτό τον άδειλο, κρυφό, αδιαφανή ε, μηχανισμό που ίσχυε στη χώρα μου μέχρι τώρα. Τι θέλω να πω με δύο λόγια. Δεν είμαι καμιά αρχοαυτόνομη που να υποστηρίζω την, ε, ε, που να είμαι κατά των υπηρεσιών πληροφοριών, του νόμου κτλ. Και δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια παρανομία γιατί δεν υπήρχε σχετικός νόμος. Ήταν απαραίτητο να υπάρξει στη χώρα μου, τη Γαλλία, ένα νομικό πλαίσιο που να είναι ξεκάθαρο και που να είναι προσαρμοσμένο στις ε, επιταγές των καιρών με την ε, πρώτων ε, νέων τεχνολογιών. Τέσσερα γρήγορα γρήγορα σημεία. Πρώτο, πρώτη ανησυχία. Η ισορροπία μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και ασφάλειας είναι ίδιο της δημοκρατίας. Υπάρχει ένας μεγάλος απόν στο γαλλικό κείμενο. που μας δημιουργεί μεγάλες απορίες και ερωτηματικά. Ο δικαστής που είναι αναγνωρισμένος για την ε, ανεξαρτησία του είναι ο θεματοφύλακας των ατομικών ελευθεριών λείπει, είναι ο μεγάλος απόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρεμβαίνει εδώ. Πρόκειται όμως για μία γνώμη που δεν ε, υποχρεώνει κάποιον να κάνει κάτι. Δεύτερον, πρώτον, να μου πείτε αν είναι συμβατά όλα αυτά με το άρθρο 2 της συνθήκης ε, και την ομολογία. Δεύτερο, δεύτερο οι συνάδελφοι θα μιλήσουν και αυτοί για τη διάρκεια φυλαξοδεδομένων και τη μαζική ε, συγκέντρωση δεδομένων. Είχα και άλλα τρία-τέσσερα σημεία, τέλο πάντων λέω πρώτα να σταματήσω. Αλλά θα ξαναγίνει συζήτηση, φαντάζομαι, όταν το Συνταγματικό Συμβούλιο θα έχει αποφανθεί και θα μπορούμε να αναφέρουμε και αυτά τα τελευταία. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να συντομεύετε καθένα στην παρέμβαση του, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, η κυρία Εντσφέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν με έχουν πείσει απόλυτα το επιχειρήματα της Επιτροπής ότι δεν ε, μπορούμε να σχολιάσουμε τις ε, νομοθεσίες των εθνικών κρατών μελών μέχρι ότου είναι καταστούν νόμοι. Όταν ο κ. Ορμπάν έθεσε την πρόταση για την θαντική πίνη, ε, σχολίασε και μάλιστα πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το αυτό πλέον αυτό το επιχείρημα. Απλά ίσως να μην θέλει να κάνει τέτοιες δηλώσεις δύσκολες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ύστερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέτε ότι δεν εκφέρει άποψη για τη συνταγματικότητα των εθνικών νόμων σε ό,τι αφορά τα εθνικά συντάγματα. Μα δεν ζητάμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη ζητάμε να σχολιάσει τη συμβατότητα όχι με το εθνικό σύνταγμα, αλλά με τι ευρωπαϊκέ συνθήκε, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώ ε, έχει εγκριθεί ο νόμο. Υπερνάει δικαστική έγκριση κάποιου είδου, αλλά έχει εγκριθεί. Έχετε νομική υπηρεσία, έχετε τοποθέτηση, άποψη. Θέλω να ξέρω ποια είναι. Είναι καθήκον σας που απορρέει από τις συνθήκες. Ύστερα. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων και ασφάλειας. Όχι. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν υπάρχει αντιστάθμιση. Είχαμε το ίδιο επιχείρημα για τα βασανιστήρια από τη CIA. Είχαμε πει τότε ότι θα πρέπει λίγο, λίγο, λίγο να κάνουμε πίσω. Τι να κάνουμε, δηλαδή λίγα βασανιστήρια για να έχουμε λίγη ασφαλεία. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύεται και συζητάμε τα βασανιστήρια, η σκλαβιά, η δουλεία, η ελευθερία έκφρασης. Είναι θεμελιώδη δικαιώματα, δεν σηκώνουν εκτόσεις. Το ίδιο ισχύει και με την ε, προστασία των δεδομένων αυτών. Και σας ανακοινώνω ότι θα θέσω παρόμοια ερωτήματα για ένα νόμο που πρότεινε μόλις η Ολλανδική κυβέρνηση που θα επιτρέπει στις μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν όλες τις επικοινωνίες μας στο διαδικτύο χωρίς ε, καμία κατηγορία, χωρίς ε, οποιαδήποτε απόδειξη μόνο στο λόγο της τιμής του δηλαδή θα πρέπει να τους πιστεύουμε ότι έχουν λόγο. Εύχομαι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατήρθει το κείμενο για την ευρωπαϊκή συνταγματικότητα. Προτού τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο νόμος. Το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο αποφαίνεται συχνά για τέτοιους νόμους, αλλά θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της, όπως το κάνει στην ταγωνιστική πολιτική, στις κρατικέ επιδοτήσεις. Γιατί δεν κάνει το ίδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκφράζω την απογοήτευσή μου που δεν άκουσα την άποψη της Κομισιόν. Πιστεύω ότι η προσφυγή του Συνταγματικού Συμβουλίου που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος των προτέρων ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να αποσιωπήσει κατά κάποιο τρόπο ή να εξοδετερώσει τις κριτικές που ακούγονταν μετά από πολλές πλευρές. Η προσφυγή βέβαια δεν είναι ούτε αυτόματη, ε, ούτε αφορά το κείμενο, αφορά κάποιες διατάξεις που ακούγονται μετα απο πολλες πλευρες η προσφυγη βεβαια δεν ειναι ουτε αυτοματη ουτε αφορα το κειμενο αφορα καποιες διαταξεις που επελεξαν οι βουλευτές. Και είμαι περίεργη να ακούσω ποια ε, συμβατότητα έχει αυτός ο νόμος με τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στις συνθήκες. Η ασφάλεια είναι ένα στόχος απλά αυτού του νόμου που έχει και άλλους στόχους, πρόληψη εγκληματικότητας, ε, καθώς επίσης και τα οικονομικά, τα μείζων οικονομικά ε, και μηχανικά συμφέροντα της Γαλλίας να προστατεύσει. Επιτρέπει μαζική παρακολούθηση από τα μαύρα κουτιά, να μπορούν να χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι στα μαύρα κουτιά και ανακαλύψαμε στη δέκα της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου ότι υπήρχε μαζική ε, υποκλοπή το 2006 για όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες ε, Γαλλίας εξωτερικού. καταγράφονται και αποθηκεύονται όλες οι συνομιλίες. Και το δικαίωμα, συγγνώμη, το, η προθεσμία είναι πολύ σημαντική. Για πόσο χρόνο δηλαδή μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα αυτά τα στοιχεία και από πότε μπορούν να, μπορούν να τα επεξεργαστούν, να τα εκμεταλλευτούν αυτά τα στοιχεία. Πολύ σοβαρά πλήγματα στι θεμελιώδει Ελευθερίε και δικαιώματα των Γαλλών πολιτών και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα το πει κάποια στιγμή Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο μελητής, κύριε Μπονφά. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως οι συνάδελφοι, οι Γαλλίδες ευρωβουλευτές, έχω παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά το νομοσχέδιο και την εξέλιξή του. Το ίδιο και τις τροπολογίες που το συνόδευαν, είτε στην Βουλή είτε στη Γερουσία. Οπότε να πω ευθύ εξ αρχή ότι θεωρώ ότι αυτό που ψηφίζουν οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες μιας χώρας, βουλευτές όπως εμείς, όχι ευρωβουλευτές αλλά βουλευτές και αυτοί, Ε, δείχνει ότι καταλήγουμε σε ένα κείμενο που είναι σύνθετο γιατί καλύπτει απόψεις και της αριστεράς και της δεξιάς. Καλό θα ήταν να σεβόμαστε λοιπόν την δημοκρατία μιας χώρας. Έπειτα το συνταγματικό δικαστήριο ε, στο οποίο έγινε προσφυγή σε πρώτη φάση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που αυτό το βρίσκω θετικό θα έλεγα ε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τι θα αποφανθεί αυτό δείχνει ε, Σοφή ότι μπορεί να ζητήσει και την απόσταση του κειμένου το συνταγματικό δικαστήριο έχει αυτό το δικαίωμα, αυτή την εξουσία, οπότε μπορεί να καταπίπτουν κάποια άρθρα. Το συνταγματικό δικαστήριο ε, εγγυάται τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στην Γαλλία. Είναι λοιπόν πολύ ωραία είδηση το γεγονός ότι έγινε προσφυγή σε αυτό και καλό θα ήταν να είμαστε συνετοί και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έπειτα, όπως είπε η Ναταλή Γκρισμπέκ, θα ήθελα πολύ να ε, ασχοληθούμε με την κατάσταση όπως έχει και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι έχουν πλαισιωμένες νομοθετικές διαδικασίες, όπως προτείνεται στο γαλλικό κείμενο, με μια Εθνική Επιτροπή ε, Ελέγχου που να αποτελείται από δικαστές, βουλευτές και συμβούλους του κράτους, οι οποίοι ε, στην αρχή της διαδικασίας να παρακολουθούν το τι γίνεται αλγοριθμικά και έπειτα ε, να υπάρχει παρέμβαση και του διοικητικού και του ε, ποινικού δικαστή. Υπάρχουν ε, ανησυχίες, λογικό είναι να ακούγονται. Πρώτη φορά έχουμε ένα κείμενο που προσπαθεί να βρει την ε, σωστή ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και του ελέγχου, αλλά ας περιμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για να πάρουμε θέση. Και κυρίως κοιτάζοντας τι γίνεται και στα υπόλοιπα κράτη, προτού αποφασίσουμε ότι το σύστημά μας προστατεύει τις ελευθερίες ή όχι, κατά τον ίδιο τρόπο σε τα κράτη της Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ και θα ήθελα τώρα να μιλήσω γερμανικά. Καταρχά. και ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις οι οποίες αντίκειται στο Σύνταγμα στις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις. Άρα ε, Αρμόζει ο έλεγχος. Κατά δεύτερον, η ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην αρχή της συζήτηση, την οποία διεξαγάγουμε εδώ και πολύ καιρό, πίστευα ότι πρέπει να υπάρχει. Εν μεταξύ, δεν μπορώ πλέον να σας πω ότι αντέχω αυτή τη συζήτηση. Είναι σαν να λέμε ότι σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κι αν λέμε ότι θα μπορούσε αυτό να αποφέρει πιο πολύ ασφάλεια. Ε, τι να κάνουμε, ας το αποδεχτούμε και ας δεχτούμε περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, όχι, δεν το δέχομαι και συμφωνώ με την ε, Σοφίν Φέλτα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα για την διαδικασία τώρα. Ναι, λήφθηκε στις 23-24 Ιουνίου μια απόφαση τυπικά ελέγχεται όλα καλά και ωραία αλλά η συζήτηση για την ομοθεσία αυτή δεν ξεκίνησε τον Ιούνιο, ξεκίνησε πολύ πιο πριν και πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε κατά πόσον κάποιες τέτοιες ανησυχητικές εξελίξεις δεν θα απαιτούσαν μια πιο έγκυρη επέμβαση. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά αν φοβόμαστε ότι ένα νομοσχέδιο κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και απασχολούν τόσο πολύ κόσμο αυτές οι προτάσεις, τι περιμένουμε να δούμε ότι δεν συμφωνούμε και θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή την όλη δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι σε, ποια, σε πιο πρώιμο σημείο θα πρέπει να εκφράζουμε τις απόψεις μας οι φήμες, οι κατηγορίες για το ότι συνέβη είναι ιδιαίτερω ανησυχητικέ αν όντω επαληθευτούν οι φήμε, ότι οι μυστικέ υπηρεσίες ε, ε, χωρίς πρόβλημα και χωρίς έλεγχο επιτρέπεται να συλλέγουν δεδομένα να παρακολουθούν πολίτες και δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος και διαφάνεια. Ούτε καν ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν βάση για τις ανησυχίες και καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκφράζεται σε λεπτομερές επίπεδο, αλλά και εδώ σύμφωνο με την Σοφίν Φέλτ ότι το κείμενο που αποφασίστηκε από την Γερουσία και του Εθνικού Συμβουλίου είναι επιτάπητος και εδώ διπλωματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, ίσως ναι, ενδεχομένω να υπάρχουν ανησυχίες ε, δεν υπάρχει βάση για ανησυχίε έτσι όπω έχει ο νόμο στην παρούσα φάση, ίσως να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η Άννα Γκόμε έχει τώρα το λόγο. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η συναδελφός ε, κυρία Σίπελ που είναι συντονίστρια της ομάδας μας. Και εγώ ανησυχώ. Και ανησυχώ και δεν αποδέχομαι το επιχείρημα από μια τέτοιες ε, δημοκρατικές αρχές. Έχω δει και άλλες δημοκρατικές αρχές από άλλες ε, δημοκρατικές χώρες να παίρνουν αποφάσεις ε, πολύ αντιπαραγωγικές και λανθασμένες σε ό,τι αφορά τα, δικαιώματα του ανθρώπου και σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας. Και εδώ αναφέρομαι για παράδειγμα στα μέτρα που έλαβε το Αμερικανικό Κογκρέσο Δημοκρατικός θεσμός τον αντιλαγεί κανείς όταν υπήρχε το πρόγραμμα των εκδόσεων ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα βασανιστήριων, τα Patriot Act και ούτω Δεν Κανεί δεν τη λέγει ότι πρόκειται για δημοκρατική χώρα. Εδώ όμως προκύπτει ότι έχουν διαπράξει σοβαρά σφάλματα. Εδώ όμως, δεδομένων των γεγονότων, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση η οποία μπορεί να αποδειχθεί πολύ παράλογη. Δεν μου αρέσουν λοιπόν αυτά που διαπιστώνω και μάλιστα από μια κυβέρνηση σοσιαλιστική της δικής μου οικογένειας που δίνει παράδειγμα, αποτελεί υπόδειγμα ε, στην Ευρώπη, είτε το θέλει είτε όχι. Άρα εδώ θα ήθελα να πω, ελπίζω να κάνει ό,τι έχει να κάνει το... το συνταγματικό δικαστήριο, αλλά ότι πρόκειται για κάτι πολύ αντιπαραγωγικό και παράλογο στον τομέα της ασφάλειας. Το τονίζω αυτό πέρα από τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που ενδεχομένω να έχουν λάβει χώρα Δεν μ' αρέσουν και αυτά που βλέπετε με τη μίλια. Και αυτά εντάσσονται λοιπόν όλα σε ένα πλαίσιο και σχετίζονται το ένα με το άλλο. Δεν μ' αρέσουν ε, τα λόγια του, Πρωθυπουργού, ε, του Γάλλου Πρωθυπουργού για ένα σοκ ε, των πολιτισμών. Ανησυχώ και νομίζω ότι οφείλω να μιλήσω ιδιαίτερα όταν βλέπουμε καταστάσεις τέτοιες καθώς πρόκειται και για μέλος της πολιτικής μας οικογένειας που διαπράττει μεγάλα σφάλματα. Thank you. Uh, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Εντφέλτ. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να δευτερολογήσω, Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια, γιατί μου προκάλεσε έκπληξη η συνάδελφο που είπε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατική απόφαση ενό ε, Εθνικού Κοινοβουλίου. Ε, ασφαλώς, αλλά ε, δεσμεύονται και από την Ευρωπαϊκό και τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Και ελπίζω να καταλάβετε την ηρωνία στο σχόλιο μου. Υπάρχει μία πόλη στη Γαλλική επικράτη την οποία θα ε, ε, επισκεφτούμε την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι θα μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος θέλετε να απαντήσετε. Και άλλο σύντομο σχόλιο. Ναι, αλλά παρακαλώ πολύ πολύ σύντομο. Να διευκρινίσω ότι φαντάζομαι ότι διάβασες το κείμενο και βλέπεις ότι έχεις δει ότι εξαιρούνται οι βουλευτές. Οι δημοσιογράφοι. Να σου α, πω όλη τη λίστα των όσων δεν συμπεριλαμβάνονται. Les avocats, les journalistes δικηγόροι, δημοσιογράφοι, δικαστές, βουλευτές, εντάξει. Απλώς για να ξέρουμε τι λέμε για το Στρασβούργο για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που δεν, Αυτό που δεν έχετε συμπεριληφθεί, ότι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι βουλευτές ε, μιλάνε με άτομα στο εξωτερικό και όταν μιλάνε με άτομα στο εξωτερικό, ό,τι λένε ε, μπορεί να υποκλέπτεται. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ψέματα της νομοστασίας αυτής που δεν έχει συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μωρίο, έχει το λόγο για να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομο. Εδώ από την αρχή φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και στο τέλος της συζήτησης το ίδιο ισχύει μπορούμε να μην έχουμε τις ίδιες απόψεις αλλά δεν μπορούμε να ε, ισχυριστούμε ότι δεν το παίρνουμε αυτό το θέμα σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην κυρία Κρισπέκ, η Επιτροπή να γνωρίζει στόματος Προέδρου της ότι ο νόμος αυτός θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα νομικά Δύο όμως ως θεματοφύλακες της συνθήκης έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία σε ισχύ ε, για την οποία να αποφανθεί η Επιτροπή και με τρόπο επίσημο. Ε, κυρία Ίντβελτ, όταν η Επιτροπή θα αποφανθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τουλάχιστον δύο κανονισμοί με το ΤΟΥΠΑΚ θα δίνουν νομική βάση για να γίνουν όλα αυτά. Ε, να γνωρίζετε, να έχετε υπόψη ότι το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το χαρακτηρίζει αυτό. Λέει η Ένωση σέβεται τις ε, κρατικές αρμοδιότητες και την ε, προστασία της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή υπερέχουν εθνικοί νόμοι για την προστασία των δεδομένων, βάσει του άρθρου 4. Βεβαίω δεν είναι βίβλο αυτό, δεν είναι δίκαιο που ισχύει θρησκευτικά, αλλά ω θρησκεία, αλλά πιστεύουμε, πιστεύω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε μια τακτική διαδικασία και ως προς το δίκαιο, νομίζω ότι όπως είπατε ο σκοπός είναι να αποφανθούμε επί της ουσίας. Δεν θα περιμένουμε 30 ημέρες του συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τα λάβει αυτά υπόψη. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και περνάμε στο Επόμενο θέμα, πρόταση για την υποφάση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη τη τρομοκρατία και του πρόσθετου πρωτοκόλου της 9 Μαου 2015. Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν ένα πρόσθετο πρωτόκολλο για την ε, σύμβαση που σχετίζεται με τους αλλοδαπούς μαχητές. Το πρωτόκολλο αυτό έχει ως σκοπό να εφαρμόσει τις πτυχές ποινικού δικαίου του 2178 για τις απειλές στην ε, ασφάλεια και την ειρήνη. Το 2015 λοιπόν ε, ενέκρινε μια απόφαση ξεκινώντας διαπραγματεύσει το πρωτόκολλο αυτό και απευθυνόμενο άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν διαπραγματεύσεις και συζητήσεις στην Επιτροπή μας και τα μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη πληροφοριών για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Και αποφάσισαν οι συντονιστές να αποσταθεί επιστολή στον κύριο Αβραμόπουλο από τον κύριο Μωράες στις 11 ε, για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μωράες όμως δεν έχει ακόμα λάβει σήμερα απάντηση. 15 Ιουνίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο αποφάσεις για αποφάσεις του Συμβουλίου για να εγκριθεί η υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σύμβασης για την Πρόληψη της Δημοκρατίας και του Προσθέτου Πρωτοκόλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εκπροσωπεί ο επικεφαλής της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ για να μας κάνει μια παρουσίαση και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψε Ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Ήμουν εδώ την 1η Απριλίου για να ενημερώσω την Επιτροπή για το πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις ανεξελίξεις τότε διαπραγματεύσεις για το πρόσθετο πρωτόκολλο και όντως λάβαμε την επιστολή του κ. Μωράης και θα πρέπει να διευκρινίσω ότι προετοιμάστηκε μια απαντατική επιστολή η οποία όμως στη συνέχεια δεν απεστάλλει γιατί είχαμε επαφές με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου της δικής μας υπηρεσίας και της Λετωνικής Προεδρίας και της επερχόμενης Προεδρίας και Έγινε μια πρώτη συνάντηση πριν από κάποιες ημέρες με τη Νέα Προεδρία και γι' αυτό θεωρήσαμε πιο σωστό και πιο αρμόζον πρώτα να σας κάνουμε μια ενημέρωση και μετά να σας στείλουμε την απάντησή σας. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο ψήφισμα του προεσμένου Σεπτεμβρίου ζήτησε από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να ποινικοποιήσουν κάποιες συμπεριφορές ε, όπως ε, η εκπαίδευση, η παροχή εκπαίδευση, σχετικά ταξίδια. Και ξέρετε ότι εκ παραλίλου, αυτό δεν ήταν καινούριο, οι ηγέτες μας ε, στο Συμβούλιο και οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών μας είχαν ζητήσει από εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουμε μία απόφαση πλαίσια του 2008 που ορίζει την τρομοκρατία. Και προβλέπει κάποιες ελάχιστες κυρώσεις. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονταν ε, εν εξελίξη το γεγονός ότι το ίσις ε, ανακήρυξε το χαλιφάτο τον Ιούνιο ασφαλώς ε, έχει μια σημασία να βρισκόμαστε σε πολιτικό κενό. Άρα στις 30 Αυγούστου του περασμένου έτους οι αρχοί κρατών είπαν να εφαρμοστεί η να, ξα... να εξεταστεί η συνθήκη πλαίσιο σε ό,τι αφορά και την ε, δικαστική απόφαση. Μετά ακολουθεί το ψήφισμα του ΟΗΕ όλο όλος ιδίω και εδώ έπαιξαν ρόλο νομίζω οι επιθέσει στο Παρίσι. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη αποφάσισε να ξεκινήσουν ε, σχεδόν άμεσα διαπραγματεύσει ε, στο πρόσθετο πρωτοκόλλο 196 για τους αλλαταπούς μαχητές. Θα θυμάστε ότι και αυτά που παρουσίασα στα κρατημέλη και εδώ Αφενός ε, κάνουμε διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα θέματα περιεχομένου, γιατί θέλαμε να αποτυπώνονται οι δικέ μα απόψει και τα δικέ μα αρχέ στο προσθέτω πρωτόκολλο. Ενώ παράλληλα κάναμε διαπραγματεύσει και εδώ στι Βρυξέλλε για εντολή. Τα γεγονότα, όπω σα είπα και τότε, δεν οφείλονται σε εμά, ε, αλλά παρόλα αυτά κληθήκαμε να τα διαχειριστούμε και θεωρούσαμε ότι ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να δώσουν όλο τους το βάρος στις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι αυτό θα σήμαινε μια κάπως ε, άμβολη διαδικασία. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις τεχνικά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέτασε το κείμενο και ζήτησε πιο πολλές εγγυήσεις, πιο πολλές ε, αναφορές και δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα έχουν προσθεθεί στο κείμενο πλέον. Και θα αναπτύξω περαιτέρω τα σχετικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι υπουργοί συναντήθηκαν εδώ στις 19 Μαΐου στις Βρυξέλλες και πολιτικά ενέκριναν το κείμενο και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της επίσημης υπογραφής και ολοκλήρωσης. Τα δύο κείμενα που έχετε μπροστά σας είναι λίγο ασυνήθιστα και αυτό γιατί, γιατί συγγνώμη, υπονομικούς όρους υπογραφή μια διεθνού συμφωνή, ενό πρόσθετου πρωτοκόλου στη συγκεκριμένη φάση. Κανονικά σημαίνει ότι τεχνικό πώ συμφωνεί κανεί με το κείμενο και ότι πολιτικό πώ προτίθεται να το εγκρίνει και να το εφαρμόσει και ότι δεσμεύεται κανείς να μην, να μην κάνει οτιδήποτε που θα διακυβεύσει την εφαρμογή του πρωτοκόλου στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι ακόμα νομικός δεσμευτικό. Νομικός δεσμεύεται μια οργάνωση ή ένα κράτος όταν το επικυρώσει. Αυτή είναι η φάση της οριστικοποίησης, της ε, ολοκλήρωσης. Αυτό πώς γίνεται συνήθως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο υπογραφών και υπογραφών και ε, ολοκλήρωσης ε, εκ Αυτό δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση όπως σας είπα και όπως συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη στη φάση της διαπραγμάτευσης, χρειαζόταν μια πιο ήρεμη και ενημερωμένη συζήτηση για τις αρμοδιότητες. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν τώρα. Οι δύο προτάσεις που έχετε πλέον μπροστά σας προκύπτουν από την ερμηνεία μας αυτή ότι για την υπογραφή της σύμβαση, συγγνώμη, πρώτα θα πρέπει να υπογράψουμε την αρχική σύμβαση. Το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου το διευκρινίζει αυτό. Είναι νομική προδιαγραφή. Δεν μπορεί κανείς να καταστεί μέλος της, του πρωτοκόλλου αν δεν είναι μέρος της σύμβασης. Εμείς δεν είμαστε προς το παρόν. Αυτό είναι νομική λοιπόν προϋπόθεση. Εδώ λοιπόν το θέμα της αρμοδιότητας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όλοι συμφωνούν ότι στην βασική σύμβαση για την τρομοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι αρμοδιότητες είναι μεικτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες αρμοδιότητες είναι κοινέ, κάποιες ενδεχομένως να είναι αποκλειστικές. Δεν έχει όμως σημασία γιατί τα κράτη-μέλη όλα, εκτός από τη Τσεχία, εκτός από τη Τσεχική Δημοκρατία, είναι μέρη της σύμβασης. Και η δική μας ε, συμμετοχή, υπογραφή και ολοκλήρωση της ε, συνθήκης θα είναι έτσι. Το βασικό και το μεγάλο ερώτημα είναι το πρωτόκολλο. Ποιος θα υπογράψει εξ ονόματος της Ένωσης, τα κράτη-μέλη, το καθένα ξεχωριστά ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Γιατί σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία και το άρθρο 3.2 της συνθήκης, πιο σημαντικό αυτό, αναφέρεται ότι υπάρχει ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη διεθνών συμβάσεων όταν υπάρχει η δυνατότητα να επηρεαστούν οι υφιστάμενοι νόμοι, η υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό ισχύει γιατί έχουμε την απόφαση πλαίσιο και άλλα νομικά εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και γι' αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ασκήσει αρμοδιότητα εσωτερικά, άρα είναι λογικό και ευλογό οι ερμές να ασκηθούν και εξωτερικά της Ένωσης σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης στην προκειμένη περίπτωση για θέματα περιεχομένου τώρα. Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο. Ουσιαστικά ποινικοποιεί πέντε συμπεριφορές. συμπεριφορές συμμετοχή σε μία οργάνωση, σε μία ομάδα που έχει σκοπό α, διεξαγωγής τρομοκρατικών επιθέσεων ή με σκοπό την τρομοκρατία, συμμετοχή άρα. Δεύτερον, ποινικοποίηση της ε, παθητικής ε, εκπαίδευσης, ποινικοποίηση ταξιδίου στο εξωτερικό για, τέτοιες, για τρομοκρατικούς σκοπούς, ποινικοποίηση της χρηματοδότησης ε, τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και η διευκόλυνση των ε, τέτοιων τρομοκρατικών ε, ε, αντικειμάτων. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν χρειάζεται τα κράτη-μέλη όταν θα μεταφέρουν τις συνθήκες αυτές, τις διατάξεις αυτές, το εθνικό δίκαιο. Εάν θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι έχουν ήδη επαρκή νομικά εργαλεία για να τιμωρούν ποινικά αυτές τις συμπεριφορές, δεν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη να επιβάλλουν ξεχωριστές, να δημιουργήσουν ξεχωριστά τέτοια τρομοκρατικά εγκλήματα. Δεν χρειάζεται να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν και να επανεφεύρουν τον τροχό. Όλες αυτές οι συμπεριφορές κατά δεύτερον, αυτές οι πέντε συμπεριφορές που σας ανέφερα θα πρέπει να είναι παράνομες και ηθελημένες. Για παράδειγμα, έστω ότι είμαι εγώ ένας τραπεζίτης. Και έρχεται κάποιος... Ε, αυτό είναι πραγματικό περιστατικό που σας αναφέρω. Πραγματική υπόθεση. Πραγματική υπόθεση και ζητώ ένα προσωπικό δάνειο 5-8 ευρώ για να ε, φτιάξω την κουζίνα μου. Υποτίθεται ο τραπεζίτης στην προκειμένη περίπτωση δρά σύμφωνα με τον νόμο και ε, προφανώς χωρίς δόλο. Δεν έχει σκοπό να, τρομοκρα... να ασκήσει τρομοκρατική ενέργεια. Απλά παραπλανάτε. Σας δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα για το παράνομο της διαδικασίας και το δόλο που θα πρέπει να υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ε, ασφαλιστικέ δικλείδε και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα, υπάρχει, θα βρείτε και στην εισαγωγή στο προήμιο σχετικέ αναφορέ και στο άρθρο 8 από πλευρά νομική δεν χρειάζονταν αυτέ οι δικλείδε, γιατί όλε οι δικλείδε τη βασική ε, σύμβαση αυτόματα ισχύουν για το πρόσθετο πρωτόκολλο. Ωστόσο, όλα τα μέρη της διαπραγμάτευσης και η συνέλευση αποφάσισαν ότι ήθελαν να επαναλάβουν κάποιες από τις δικλείδες αυτές. Ως εκ τούτου αυτές οι αναφορές είναι στο προημείο και στο άρθρο 8 όπως σας είπα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας απόλυτα. Κατά δεύτερον, ότι χρειάζεται εγγύηση του δικαιώματος σε ότι το βάρος απόδειξης είναι τον κατηγορό, στον εισαγγελέα και δεν ε, βαρύνει τον κατηγορούμενο. Και ασφαλώς ε, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της αθωότητας ε, σε όλες τις περιπτώσεις. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, που βρισκόμαστε λοιπόν στην παρούσα φάση με τη βοήθεια της επερχόμενης Προεδρίας, της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, πριν από κάποιες μέρε έγινε μια πρώτη απόπειρα, μια πρώτη συνεδρίαση και ε, προγραμματίζονται άλλε τρει συναντήσεις μέσα στον Ιούλιο για να διευκρινίσουμε το θέμα της αρμοδιότητας. Έχουν αποκλίνει στις απόψεις τα κρατημέλη επ' αυτού. Η Τσεχική Δημοκρατία ε, έχει πρόθεση να επικυρώσει την βασική σύμβαση. Αυτό είναι στα δικά της χέρια πλέον. Και αν υπάρχει νομίζω σχετική ορμή στην πράγμα, σχετική κίνηση για να, να αναλυφθούν οι κατάλληλε δράσει, κάποια κρατημέλη θεωρούν ότι το σύνολο ή κάποιο τμήμα του πρωτοκόλλου αποτελεί κοινή αρμοδιότητα. Εδώ διαφωνούμε. Πρόκειται για την νομική ερμηνεία της ε, συνθήκης και της σχετικής νομολογίας. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και θα ήθελα να σα το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, στον κύριο Βέμπερ από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου. Σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Που δίδεται συγκεκριμένα στην Προεδρία του Λουξεμβούργου το λόγο. Για να πει κάποια λόγια και αυτή την πρόταση απόφασης. Ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό σας τα εξήγησε ήδη. Έχουμε δύο προτάσεις λοιπόν σε σχέση με το το πρωτόκολλο, η πρόταση απόφαση υπογραφή τη σύμβαση εκπήρες από την ανάγκη να είμαστε μέλη της σύμβασης της αρχής για να μπορούμε να ενταχθούμε και στο πρωτόκολλο. Το συμπληρωματικό, ξέρουμε πώς γεννήθηκε αυτό το πρωτόκολλο, τα είπε και ο εκπρόσωπος ε, της Κομισιόν και εξήγησε και την κάπως ασυνήθιστη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου σε ό,τι αφορά τις εργασίες για τις δύο προτάσεις σε επίπεδο Συμβουλίου τα κράτη-μέλη είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις αρχές της ε, εβδομάδας αυτής ακόμη επί Λετωνικής Προεδρίας η Λουξεμβουργιανή Προεδρία προβλέπει τρεις συνεδριάσεις εντός του Ιουλίου με στόχο έγκριση κατά το φθινόπωρο και επί της ουσίας νομίζω ότι ο πρόσωπος Επιτροπής πολύ καλά εξήγησε που είναι ε, τα σημεία αποκλήσεως μεταξύ της άποψης της Κομισιόν και της πλειοψηφίας των κρατών μελών του Συμβουλίου. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα παρακαλώ όποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Ντεπχέ καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχα άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Άρα έχασα ένα μεγάλο μέρος της παρέμβασής σας, οπότε ίσως να, μην, να είμαι εκτός θέματος. Και να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Δεν θα μιλήσω επί της ουσίας, γιατί συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την ουσία, αλλά για τη διαδικασία θα ήθελα να μιλήσω. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο, θα πρέπει να υπογράψουμε καταρχάς τη σύμβαση, την αρχική σύμβαση. Πόσα κράτη έχουν ήδη από το Συμβουλίο της Ευρώπης ε, υπογράψει αυτή τη σύμβαση, για να έχουμε μια ιδέα του αριθμού του πόσοι μπορεί να ενταχθούν και στο πρόσθετο πρωτόκολλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπογραφή του του πρωτοκόλλου. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι με βάση την ανάλυση του άρθρου 3.2 της ε, συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία πρέπει να προσυπογράψει αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο. Έτσι δεν είπατε. Ωραία. Σας πιστεύω, αλλά διαβάζω και τον τύπο. Για δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί ε, το πράγμα. Για το σημείο 4 λέγεται ότι κάθε πλευρά εγκρίνει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να επιβάλλει ποινικέ κυρώσει θέματα ποινικού δικαιώμα. Δεν έχουμε εμεί ω Ένωση αρμόδια σε θέματα ποινικά, άρα πώ μπορούμε να υπογράψουμε δεσμεύοντα αυτού που δεν είναι ε, συμβαλόμενα μέρη και θα πρέπει να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο κάποιε διατάξει, γιατί αυτό το βλέπουμε σε κάθε άρθρο. Για όλε τι ε, παραβάσεις που θα ε, διαπιστωθούν. Άρα υπάρχει ένα ενοιολογικό πρόβλημα. Αν μπορείτε να μου το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί τέλειο υποσύγχυση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελα να λάβει το λόγο, να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Λούς για να απαντήσει. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ για να σας ε, διαφωτίσω. Στο πρώτο σας ερώτημα η απάντηση είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την Τσεχική Δημοκρατία όχι απλά έχουν υπογράψει αλλά και έχουν επικυρώσει την ε, σύμβαση. Άρα είναι συμβαλόμενα μέρη από νομικής πλευράς αυτής της σύμβασης. Όπως είπε η Λουξεμβριανή Προεδρία, αυτό είναι προαπαιτούμενο επιβάλλεται από το πρωτόκολλο. Δεν μπορεί, ε, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, να μπορεί κανεί να είναι συμβαλόμενο μέρο του πρωτόκολλου και όχι τη σύμβαση, που είναι το αρχικό νομικό έγγραφο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε, ξέχασα να σα πω ότι είναι το άρθρο 3.2 ε, τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το άρθρο λοιπόν προβλέπει, ορίζει ένα κλειστό κατάλογο αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης και υπάρχει και το εδάφιο 2, δεν το έχω μπροστά μου βέβαια, που λέει ότι υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα επίσης όταν η σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του πεδίου εφαρμογή των κανόνων των ευρωπαϊκών που ισχύουν. Και εδώ έχουμε ε, την απόφαση πλαίσιο από το 2002 που αναθεωρήθηκε το 2008. Άρα την έχει την αρμοδιότητα η Ένωση και το 2002 και το 2008 την έχει διασκήσει. Και ήμασταν τότε στον τρίτο πυλώνα. Ήταν αποφάσεις πλαίσια και όχι κανονισμοί ή οδηγίες. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, από την αρχή πριν τα δραματικά γεγονότα του Παρισιού και πριν το Συμβούλιο της Ευρώπης δεσμευτεί πάρα πολύ γρήγορα και κάπως έτσι με αυτοσχεδιάζοντας ε, μας έβασε μια δύσκολη διαδικασία. Είχαμε την εντολή να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την λισαβονοποίηση, μου επιτρέπετε, της απόφασης πλαισίου. Όχι δηλαδή απλά να ξανασυζητηθεί το περιεχόμενο, ώστε ακριβώς να απαντήσουμε ή να ανταποκριθούμε σε αυτό το φαινόμενο των ε, ξένων μαχητών και να δώσουμε και μια πολιτική απάντηση και Συμβούλιο ασφάλιση των Εθνών, αλλά ήθελα ε, μεταφορά, επειδή δεν υπάρχει τρίτο πυλώνα, ε, στον πρώτο πυλώνα, να κοινοτικοποιηθεί ε, αυτή η απόφαση πλαίσιο. Και αυτό έχει κάποια νομικά και έχει κάποιες νομικές συνέπειες επί της ουσίας τώρα. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι λάβαμε την εντολή από τα κρατη από τους αρχηγούς καθών και κυβερνήσεων, να αναθεωρήσουμε αυτή την απόφαση πλαίσιο. Άρα υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο που έχουμε στη διάθεσή μας και πρόθεσή μας είναι, όπως υπόθηκε και στο νέο θεματολόγιο για την ασφάλεια, άρα έχει επικυρωθεί στο ύψιστο επίπεδο από την Κομισιόν. Δεν σα το λέει ένα απλό υπάλληλο, ο Σώμα των Επιτρόπων το αποφάσισε. Για το 2016, οι παρασκευαστικέ εργασίε έχουν ξεκινήσει. Άρα, θέση μα είναι ότι είμαστε στην ε, κατηγορία ε, που προβλέπεται στο άρθρο 2, 3, δάφιο 2 τη Συνδίκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρμοδιότητα και μπορούμε να προβλέψουμε αλλαγή. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη και το εν λόγω πρωτόκολλο έχουν επίπτωση συγκεκριμένη στην νομοθεσία. Και να πω, απαντώντα στο τελευταίο σα ερώτημα, ότι κάθε συμβαλόμενο μέρο καλείται να εφαρμόσει αυτό το πρωτόκολλο. Φυσικά, δική μα πρόθεση είναι να προτείνουμε ευρωπαϊκού επίπεδου εναρμονισμένη εφαρμογή με αυτήν την οδηγία. Για κάποια κράτη-μέλη δεν θα έχει νόημα, αφόσον έχουν ήδη τα σχετικά νομικά μέσα. Για κάποια κράτη δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή, αλλά για άλλα κράτη αλλαγές υπάρχουν. Γιατί θα πρέπει να τροποποιήσουν ε, την, ε, τον ποινικό χαρακτηρισμό ορισμένων από τις παραβάσεις που ανέφερα και να κάνουν σχετικές αλλαγές στο Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πέρα από τη διαφωνία ως προς τις αρμοδιότητες, τις νομικές αρμοδιότητες ας πούμε, τι θα ήταν πιο γρήγορο και πιο σύμφωνο με τη φιλοσοφία καταπολέμησης της τρομοκρατίας αλλά και το σεβασμό των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί της ουσίας, τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν προς το πρωτόκολλο. Αυτό πρέπει να γίνει και σε υπουργικό επίπεδο πέρασε αυτό το θέμα. Υπάρχει συμφωνία από το λοιπόν από πολιτική άποψη αλλά και νομικά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει διαδικασία υπογραφή και μετά ε, ολοκλήρωσης και κυρώσεις. Όπως είπα στην αρχική μου εισηγήση. Είναι δύο ξεχωριστά κείμενα, αλλά συνήθω ε, προτείνονται ταυτόχρονα εδώ για σκοπούς σωστής διαλέγγανσης τη υπόθεση προτάθηκε να γίνει διέρευση του πακέτου με δύο αποφάσεις προς και το φθινόπωρο δύο προτάσεις συμπρασμάτων ελπίζω. Αν παραμείνουμε στη θέση ότι η διαδικασία είναι μεκτή, η κύρωση θα αργήσει. Διότι και η Ένωση και καθένα από τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσει το πρωτόκολλο και η διαδικασία κυρίω πρέπει να γίνει ξεχωριστά με διαφορετικού ρυθμούς, επειδή ο καθένα έχει τη δική του χώρια διαδικασία που διαφέρει. Εάν όμω ακολουθήσουμε το κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία της αποκλειστικής αρμοδιότητας. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιστότερη στο πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντεπρέ, να είμαι βέβαιος ότι σωστά κατάλαβα. Όταν το άρθρο 4-5 λέει ότι κάθε μέρος θα χρησιμοποιείται διάταξη που φαίνεται κατάλληλη για την ποινική παράμβαση. Θα πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποια οδηγία θα καλεί τα κάτι μέλη να προκλέψουν στο ποινικό τους δίκαιο τις, τα δικήματα που, διαβάζονται, που απαριθμόνται εδώ, με το είδο κυρώσεων που θα πρέπει να αντιστοιχούν. Αυτό είπατε ακριβώ. αρχίζω να γίνομαι όλο και πιο καχύποπτο. Uh, uh, Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Να συνεχίσουμε να περιμένουμε. Um, Το επόμενο θέμα είναι παρουσίαση της νομοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου γιατί τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 οι συντονιστές αποφάσισαν την απλουστευμένη διαδικασία βάσει του, κανόν, του άρθρου 50 του εσωτερικού κανονισμού για την έγκριση της θέσης του Ευρωκοινοβουλίου για τις τρεις αυτές υποθέσεις. Μιλάμε για τρεις εκθέσεις με εισηγητή και στις τρεις περιπτώσεις τον Κλοντ Μωράης. Στην συνεδρίαση ΛΥΜΠ 14 Απριλίου 2015 το Συμβούλιο μας ενημέρωσε ότι προβλέπει αρκετέ αλλαγέ στην πρόταση τη Επιτροπή και υπεύρεται τι βασικέ του τροπολογίες. Η Επιτροπή συμφώνησε στι τροπολογίε του Συμβουλίου και βάσει των τροπολογιών του Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2015 οι συντονιστές αποφάσισαν να ε, ζητήσουν από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου γνωμοδότηση για τα τρία αυτά θέματα, ιδίω για τις πιο σημαντικές τροπολογίες που πρότεινε το Συμβούλιο. Η γνωμοδοτήση απεστάλλει στον κύριο Μωράη στις 23 Ιουνίου και μοιράστηκε σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΑ. Κατά πρώτον να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Υπάρχουν τρει προτάσει τη επιτροπή, Επιτάπτως για συζήτηση από την Επιτροπή σα, Κάθε μια από αυτέ βασίζεται σε διάφορε νομικέ βάσει και σκοπό έχει να ανακαλέσει διάφορε παροχημένε πράξει στον τομέα τη ελευθερία, ασφάλειας και δικαιοσύνη. Η νομική υπηρεσία έλαβε δύο ερωτήσει από τη δική σα πλευρά σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν η επιλογή κανονισμού ω είδο πράξη για του σκοπού αυτών των τριών προτάσεων συνάδει με τις συνθήκες. Απαντήσαμε στην ερώτηση αυτή καταφατικά και για τις τρεις προτάσεις. Ένας κανονισμός είναι η καταλληλότερη επιλογή, η σκοπιμότερη επιλογή και για τις τρεις προτάσεις. Καταρχάς, να υπογραμμίσω ότι η συνθήκη δεν επιτρέπει ιδιαίτερο είδος πράξης να χρησιμοποιείται για την ανάκληση πράξεων της Ένωσης. Απλώς λέει ότι αν η συνθήκη δεν διευκρινίζει τι είδος πράξης πρέπει να επιλογεί, οι θεσμικά όργανα μπορούν να επιλέγουν περίπτωση. Υπάρχουν δύο προτάσει, οι νομικέ βάσεις που προτείνονται από την Επιτροπή, να μην διευκρινίζει το είδο πράξη που θα προτιμάτε. Αυτέ οι νομικέ βάσει αναφέρονται απλά και ασαφώς και γενικά σε μέτρα εντό εισαγωγικών. Γι' αυτό, για την περίπτωση αυτών των προτάσεων, θα δώσω του αριθμού τη σειρά του COM 2014-713 και 714, σε αυτές τις περιπτώσεις το σώμα καταρχήν είναι ελεύθερο να επιλέξει την καταλληλότερη μορφή πράξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθεί η απόφαση για την ανάγκηση των πράξεων αυτών. Σύμφωνα με το σχέδιο του Συμβουλίου, το Συμβουλίο θεωρεί ότι το είδος του εργαλείου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ο κανονισμός. Μελετήσαμε το αν υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ του κανονισμού της απόφασης για τις προτάσεις αυτές ε, κοιτάξαμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει το τελικό αποτέλεσμα μιας απόφασης μπορεί να είναι το ίδιο όπως αυτό μιας άμεσα εφαρμόσιμης διάταξης κανονισμού. Ιδίω αν η διάταξη δεν περιλαμβάνει προποθέσει και είναι αρκετά σαφή και ακριβής. και ακριβής. Βάσει της δικής μας εξέτασης, μια απλή ανάκληση ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα απόφασης κανονισμού είναι παρόμοια. Διαφέρει κάπω η περίπτωση της τρίτης πρότασης της Επιτροπής ΚΟΜ 2014-715. Δύο από τις νομικές βάσεις της τρίτης πρότασης διευκρινίζουν τι είδου πράξεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το άρθρο 83.1 της συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει καταρχήν την έγκριση οδηγιών και το άρθρο 88.2 της συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την έγκριση κανονισμών. Και η, Προ... Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν ότι ο κανονισμό είναι σκοπιμότερο για την τρίτη πρόταση. Ο κανονισμό είναι το ίδιο εργαλείο που συνάδει με όλε τι νομικέ βάσει τη πρόταση. Επιπλέον, ε, το να ανατρέξουμε σε κανονισμό απαιτείται και από το άρθρο 88.2, μια από τι νομικέ βάσει. Ο κανονισμό λοιπόν είναι το σκοπιμότερο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί για την τρίτη πρόταση. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναλύσω το θέμα του άρθρου 83.1. Αυτή είναι μια από τις νομικές βάσεις της τρίτης πρότασης. Απαιτεί την χρήση οδηγιών σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων. Ωστόσο, η νομική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η καταγράμμα ερμηνεία της συνθήκης δεν είναι η μόνη δυνατή επιλογή. Επειδή ο στόχος της πρότασης δεν είναι η έγκριση νέων μέτρων εναρμόνισης, αλλά απλώς η ανάκληση ξεπερασμένων πράξεων, η χρήση και το να τρέξουμε σε οδηγία δεν φαίνεται να είναι κάτι που απαιτείται. Στο δεύτερο τμήμα της πρώτης σας ερώτησης, ρωτήσατε εάν υπάρχουν νομικά επιχειρήματα υπέρ του να επιλογεί κανονισμός αντί για απόφαση. Όπως είχα αναφέρει στο παρελθόν, μάλλον όπως ανέφερα νωρίτερα, η ερώτηση αυτή αφορά μόνο τη δεύτερη και την πρώτη πρόταση, αλλά το σώμα δεν υποχρεούται να προτιμήσει τη μια την άλλη μορφή πράξης. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα απόφαση ή κανονισμού ε, είναι παρόμοια για την περίπτωση ανάκλησης τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, η νομική μα υπηρεσία δεν βρήκε κάποιο ε, ε, Κάποια διαμφισβήτη το επιχείρημα υπέρ της μιας της άλλης λύσης. Για τη δεύτερη ερώτηση θεωρούμε ότι το, το Συμβούλιο θεωρεί μάλλον ότι η απόφαση πλαίσιο είναι η καταλληλότερη περίπτωση για την ανάκληση. Ε, χρειάζονται μεταβατικέ διατάξει και τροπολογίε σε κάποιε συλλογικέ σκέψει για αυτή την επιπλέον ανάκληση. Να θυμίσουμε ότι η απόφαση πλαίσιο έχει ήδη αντικατασταθεί από την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη σε ποινικέ υποθέσει. Αυτή η οδηγία θα ισχύσει και για τα 26 κράτη-μέλη, με την εξαίρεση τη Δανία και τη Ισλανδία που δεν συμμετείχαν στην έγκρισή τη. Η νομική υπηρεσία εξέτασε τι προτινόμενε διατάξει και το νομικό πλαίσιο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάκληση τη απόφαση πλαισίου για το Ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων δεν εγείρει νομικέ ανησυχίε. Όμως, και θα κλείσω με αυτή την παρατήρηση, η ευκαιρία για τέτοια ανάκληση θα πρέπει να αποτιμηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Συνάδελφοι, θέλετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, όχι. Αν όχι, ο κύριος Μωρές λέει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με βάση την απλουστευμένη διαδικασία με τροπολογίες. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ο κύριος Μωράης ως εισηγητής θα συντάξει τις προτινόμενες τροπολογίες με βάση τη συζήτηση και τις τροπολογίες του Συμβουλίου. Αυτές οι τροπολογίες σας αποσταλούν μέσω email μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και δυνάμει του κανάλι 50 θα μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση εντός προθεσμίας στις τροπολογίες, αλλιώς θα θεωρηθεί η έκθεση ότι εγκρίνεται μαζί με αυτές τις τροπολογίες και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Εάν υπάρξουν ενστάσεις, στην επόμενη συνέντευξη της ΛΥΠΑ θα ψηφιστούν αυτές τις τροπολογίες. 21 ημέρες είναι το πολύ η προθεσμία, μάλλον το λιγότερο η προθεσμία 3 Ιουλίου. Ξεκινάμε, άρα 24 Ιουλίου λίγη προθεσμία. Γιατί θέλουμε να είναι πιο σύντομη δυνατή για να προχωρήσουμε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τρεις αυτές εκθέσεις και τις νομικές γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας. Και έχουμε και άλλο ένα σημείο τελευταίο στην Μεσσιαδιάταξη, δηλαδή την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση αποστολή αντιπροσωπεία τη Λίπρα στην Ουάσιγκτον από τι 16 έω τι 19 Μαρτίου. Κεφαλή ο κύριο Άλμπρεχτ. Προετοίμασε το σχέδιο έκθεσης μαζί με τα άλλα μέλη της αποστολής που είχε ως στόχο να συγκεντρώσει επικαιροποιημένες πληροφορίες για την κατάσταση και την πρόοδο στις Πολιτείες για σημαντικά στήματα που αφορούν την προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένου μετά το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου του 2014 του Κοινόβουλου για τις μαζικές ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις PNR μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΠΑ, TTIP, συμφωνία Αμπρέλα, νομοσχέδιο για επέκταση των ε, διατάξεων και για μη Αμερικανούς υπηκούς κτλ. κτλ. Είναι να συναντήσει αρκετές με μέλη του Κογκρέσου, ΜΚΟ ε, και βέβαια και με την κυβέρνηση. Δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες και βοήθη απέκτησαν οι ανταλλαγές την καλύτερη συνεργασία με τις αρχές τη κυβέρνηση και του Κογκρέσου. Και αυτή τη συνεργασία θέλουμε να την ενισχύσουμε, να έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν αρμοδιότητες τη Επιτροπής μα, ιδιωτική ζωή, ασφάλεια, πολιτικές ελευθερίες, μεταφορά δεδομένων. Θα μπορούσαμε να διτυπώσουμε ω Λίμπε συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιος θέλει να σχολιάσει κάτι. Φαίνεται ότι είμαι η μόνη, το μόνο μέλος που μπορεί να αποδείξει ότι αυτά που λέει η έκθεση ισχύουν. Πραγματικά συνέβησαν και πραγματικά είχαν αντίκτυπο στη μελλοντική εργασία των μέλων στο, σε ό,τι αφορά διάφορα νομοθετικά πακέτα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ότι ένας από τους στόχους μας ήταν επίσης να γίνει εκτενής διάλογος με την Αμερικανική πλευρά προκειμένου να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές διαφορές και μήπως πρόκειτο όχι για πραγματικές διαφορές, αλλά για μετάφραση διαφορετικών ε, νομικών ερμηνεών, διαφορετικών ε, πολιτισμών. Και κατανοήσαμε λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις ότι το κενό δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο πιστεύαμε, ενώ αλλού διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πραγματικά προβλήματα που δεν είχαν επιλυθεί. Άρα αυτές οι άμεσες επαφές, αυτός ο διάλογος πραγματικά αποδείχθηκε πάρα πολύ και ένα συγκεκριμένο καθήκον ήταν αυτό το νομοσχέδιο το οποίο τότε είχε να κάνει με την εξίσωση των δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων πολιτών με τους Αμερικανούς. Και εδώ αντιδράσαμε πολύ διαφορετικά προκειμένου να κάνουμε να καταλάβουν ότι πραγματικά χρειαζόταν το νομοσχέδιο αυτό. Ήταν πολύ λοιπόν ε, χρήσιμη η επίσκεψη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε την συνεδρίαση αυτή. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει στο Στρασβούργο 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και γεια σας.